que hemos dado a todo el mundo para que venga aquí y yo eh, voy a empezar la votación del informe de la señora Lovín sobre la pesca yuyú. Ε, ξεκινάμε με την ε, έκθεση της κυρίας Λεβίν. Παρακαλώ καθίστε όλοι για να ξεκινήσουμε την ψηφορία. Περίπλοκη ψηφορία. είχαμε την τελευταία στιγμή προφορικές τροπολογίες και θα πρέπει να θέσουμε και κάποια προθεσμία ε, για τις προφορικές τροπολογίες. Διαφορετικά κατάσταση είναι χαόδης. Θα ξεκινήσουμε πάντως την ψηφοφορία. Έχετε όλη την κάρτα, ελπίζω. Ωραία, πολύ ωραία. En primer lugar, someto a votación Να με, ψηφίζοντας λοιπόν, τροπολογία 22. Κυρίες και κύριοι, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με νέα ψήφους. Στη συνέχεια θέτω σε ψηφοφορία τη συμβαστική πρόταση 2. Άρχεται η ψηφοφορία. 2 και 3 μαζί, συμβαστικέ προτάσει, 2 και 3 μαζί. Άρχεται η ψηφορία. Πέρα τη ψηφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτουν λοιπόν οι 15, 16, 17, 18, 19, περιβάλλοντος 5, 6, 14 και η τροπολογία 21. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συμβαστική πρόταση 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτουν 24, 25, 26, 29, 28 και 27 τροπολογίες. Θέτω σε ψηφορία τώρα την συμβαστική πρόταση 5. Άρχεται η ψηφορία. Πέρα της ψηφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτουν οι 30 και 35 τροπολογίες. Ψηφίζουμε 31. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα την τροπολογία 32. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 8 ψηφί υπέρ, 7 κατά. Τροπολογία 33 τσουκαλά αποσύρθηκε. Θέτω τώρα, όχι, η 34 καταπέπτει επειδή ακριβώς η 32 εγκρίθηκε. Συμβαστική πρόταση 6. Ψηφίζουμε. Πέρα Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Καταπίπτουν 36 και 46. Θέτω σε ψηφορία την τροπολογία 11 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 8-8 απορρίπτεται. Θέτω τώρα σε ψηφοφορία την 13 της περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. 8 υπέρ, 7 κατά, εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται ομόφωνα. Στη συνέχεια, στην 38 τροπολογία, έχουμε προφορική τροπολογία Κρίστενσεν. Έχετε το λόγο. Κύριε Κρίστενσεν, έχετε το λόγο. Κυρία Λόβιν. Ωραία. Θα προσπαθήσω να δεχτώ την προφορική τροπολογία Κρίστεσεν. Καλεί την Κομισιόν να διερευνήσει μέχρι το 2014 κατά πόσο η ψυχαγωγική αλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως IUU Fishing. Τελεία. Και διαγράφεται η υπόλοιπη τροπολογία. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Υπάρχει ένας φιλελεύθερος παραπάνω. Κύριε Γκάλαχερ, θα πρέπει να διώξετε ένα από τους ψηφοφόρου σα εδώ πέρα. εσεί που είστε συντονιστή. Bueno, την ψηφοφορία. Ξαναψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε cierra. Πέρας Εγκρίνεται. Στη συνέχεια τίθεται σε ψηφορία η τροπολογία, η προφορική 1, καντά κρυβελίνη που αντικαθιστά την 62 και 39 τροπολογία. Ένας από τους δύο να λάβει το λόγο. Δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Ωραία, θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια καταπίπτουν οι 62 και 39. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφορία, Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται Τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε θύρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 43, 44, 45 και 90. Θέτω σε ψηφορία την τροπολογία 20 περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφορία πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 11 υπέρ 8 κατά. Θέτω τώρα σε ψηφοφορία την συμβαστική πρόταση 8. Ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία εκ μέρους του ΠΠΕ. Θέτω σε ψηφοφορία το πρώτο τμήμα της τροπολογίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό. Καταπίπτουν οι 50, οι 85. Συγγνώμη λέει... Κατά λίγο ησυχία, αλλιώ μπερδεύομαι, λέει η πρόεδρο. Λοιπόν, καταπίπτουν οι 50, οι 85, οι MV7, το δεύτερο τμήμα. Οπότε θέτω σε ψηφοφορία την ε, συμβαστική 9, η, η Προφορική τροπολογία. Έχετε το λόγο. Ναι. Θα θέλαμε να πούμε το εξή. Λέει εδώ πέρα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, κατα... καταπολεμήσει την παράνομη ελεία, θέτοντα σε εφαρμογή και εφαρμόζοντα τα αντίστοιχα και απαραίτητα μέτρα, τι συμφωνίε κλπ. κλπ. που απορρέουν από το δίκαιο τη θάλασσα. Όπω επίσης και τα διάφορα προγράμματα αλλιευμάτων, όπω αυτά έχουν υιοθετηθεί διεθνώ κλπ. κλπ. Είμαστε υπέρ ως συζητητέ. Ωραία. Αν δεν διαφωνεί κάποιο, θέτουμε σε ψηφοφορία την συμβαστική 9, όπω ακριβώ τροποποιήθηκε, όπω την ακούσαμε την εισηγήτρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα καταπίπτουν οι 51, 52, 72, οι 3, οι 3 ντεβε, συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφορία. Πέρα της ψηφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτουν οι 55, 56, 57 τροπολογίες. Ψηφίζουμε για τη συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφορία. Σε Πέρας εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτουν οι 64, 48, 69 και 103 τροπολογίες ψηφίων για τις 47. Άρχεται η ψηφορία. Πέρα. Πέρας εγκρίνεται. 49. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 19 περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Περάς. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 12. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 59, 60 και 61. Θέτω σε ψηφορία την τροπολογία 58. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 63. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφορία την 1 Ανάπτυξης. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. δύο, Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία παριθμών 4 της ΔΕΒΕ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 5 της ΔΕΒΕ, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13, ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται κατά 66 και 67 και ψηφίζουμε την υπαριθμόν 53. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Την υπαριθμόν 6 της ΔΕΒΕ. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 18 και 21 της ΕΝΒΕ. Και ψηφίζουμε την 7 της ΔΕΒΕ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 68. Πατράω Νέβες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και απορρίπτεται 11.39. 70. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με χωριστή ψηφοφορία η 71. Το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Se cierra. Aprobado. Segunda Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα. cierra. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε. Είναι 73. Ψηφίζουμε. Σε cierra la votación. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 74. Ψηφίζουμε. Σε cierra. Aprobada. Someto a votación la enmienda 75. 75. Ψηφίζουμε. Σε cierra. Πέρασε. Και απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 76. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 77. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 78. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 79. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 80. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 81. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 82. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απολύτω. 83 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 84 έχει αποσυρθεί. Προφορική τροπολογία παριθμών 2. Του κυρίου Μιλάνα έχει αποσυρθεί και άρα πάμε στο 87. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 88. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 89. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ένβη. 9. Πρώτο τμήμα. Α, όχι, όχι. Έχει εγκριθεί 89 για ε, αυτή αυτή πίπτη. 92 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 14-6. Ένβη 9. Έχει και αυτή καταπέση. 91. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 93. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 95. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 94. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται. 96. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται. 97. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται. 98. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 99. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 100. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 101. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. MV10. Καταπίπτει. Προφορική υπαριθμόν 3. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 102. Έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία 4 της ΕΜΒΗ. Ψηφίζουμε. Πέρας. 12-8 εγκρίνεται. 104. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 86 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 105 ψηφίζουμε. Πέρασε. 10-10 καταπίπτει. 107 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 108. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται και καταπίπτουν οι 109, 106, 110 και η, το πρώτο τμήμα της ΕΝΒΗ 15. 111 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Καθημερινά 113, 112, 114, 115, και το πρώτο τμήμα της ΕΝΒΗ υπαριθμών 2 και ψηφίζουμε 116. Πέρασε. Εγκρίνεται. 117 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απόλυτος. 118 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 119 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 120 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται 121. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 122. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογικό παριθμών 2. Ψηφίζουμε. Σε φιέρα. Πέρασε. Απολύτω. Παριθμών 13. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απολύτως. 4. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 5. Ψηφίζουν. Πέρασε. Απολύτω. 6. Πέρασε. Απορρίπτεται 18. Τροπολογία υπαριθμών. Α, καταπίπτει 7. Κατόπιν στην υπαριθμών 8 έχουμε απόσυρση όμως έχουμε για αυτή την αιτιολογική παράγραφο μια προφορική τροπολογία του κύριου Κρίτσνεσεν ο οποίος δεν είναι εδώ άρα α εδώ είναι εδώ είναι α, καλώς τον έχετε το λόγο ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να σας διαβάσω παράνομη αλία έχει αναφερθεί μεταξύ 11 και 26 εκατομμύρια τόνων. Δηλαδή περίπου το μισό του αλίευματος. Και οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ε, παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση των παγκόσμιων πόρων. Ποιος σωστά κάνει αδύνατη τη διαχείριση των πόρων παγκοσμίω. Πέρας, λέει πρόεδρος και εγκρίνεται. Καταλαβαίνετε, η 9, 10 και ψηφίζουμε την 11. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 13, 23 και 14 καταπίπτουν. Και ψηφίζουμε το ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ομόφωνη εγκρίνεται, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Οπότε και έτσι ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερησίας Τι; Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο. Για να δεν κάνω λάθος. Τι είχαμε σήμερα, ποιο τι ήταν. Έχουμε αλλάξει τόσες φορές τη μέση διάταξη. Α, κυρία Τροτμάν, έχετε το λόγο. Ποιο ήταν, το 5. Το 5. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Σε σχέση με την γνωμοδότηση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Επιτροπή είναι επί της ουσίας πάνω σε αυτό. Από τον Ιανουάριο ασχολούμαστε με αυτό το θέμα για τη βελτίωση και την απο... σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα αποθέματα. Γίνεται μια με πολύ πλευρή, θα λέγαμε, αντιμετώπιση του θέματος, πολλές πτυχές και εγώ θα στηριχθώ σε σχέση με το παράκτημα που έχουμε, αλλά θέλω να το δω και πιο ευρέως όσον αφορά τους στόχους που θέτουμε εμείς. Τρεις είναι οι, οι, οι βασικοί άξονε, θα λέγαμε. Η διαχείριση των αποθεμάτων καταρχήν. αυτό είναι ο βασικός στόχος μας. Και πέρα από τον ορισμό των ε, αποθεμάτων, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέσα για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματικότητα, διότι εδώ υπάρχουν αντίθετε απόψει. Μετά το θέμα με την απόρριψη των αλλιευμάτων, ε, την εμπορική πτυχή και τη διεθνή διάθεση, διάσταση αυτού του θέματος. Αυτά είναι τα πρώτα μου σημεία. Μετά, το θέμα της προστασίας του οικοσυστήματος είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να παντρέψουμε ε, οικονομικές ε, ανάγκες των ψαροάδων και τις ε, οικολογικές πτυχές. Θα δουλέψουμε από κοινού για τα έγγραφα στο μέλλον. Πρώτον, τώρα, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ούτως ώστε οι αλείς να σέβονται αυτή τη διάσταση, να γίνονται σεβαστά τα ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία υπάρχουν και επίσης θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και κινητοποίηση όσον αφορά αυτή, αυτό το θέμα. Επίσης, να γίνει μια κοινή προσπάθεια όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική για να προστατευτούν τα αποθέματα. Και τρίτο θέμα τώρα θα ήθελα εγώ ε, να δω το θέμα που έχει να κάνει ε, το θέμα των καυσίμων εδώ. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ε, μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν από τη μια το περιβάλλον αλλά θα βοηθήσουν και τους αλληλείς. Θα πρέπει φυσικά θα πρέπει να δούμε και το θέμα το οποίο έχει με την απερελίευση ε, στη θάλασσα. Τώρα φυσικά έχουμε μια πρώτη παρουσίαση, αλλά θεωρώ η Επιτροπή μας θα πρέπει ε, να δώσει ένα μήνυμα στον τομέα αυτό και θα πρέπει εδώ να συνεργαστεί με τους ε, επαγγελματίες για μια βιώσιμη, θα λέγαμε, δραστηριότητα. Εδώ είναι μια λεπτή, θα λέγαμε, προσπάθεια, δραστηριότητα, είναι όντως ένα έργο το οποίο είναι σίγουρα ενδιαφέρον διότι γίνεται, θα λέγαμε είμαστε στο προστάδιο της μεταρρύθμισης που θα γίνει όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική. Αυτά προς το παρόν κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τρότμαν. Ο κύριος Βατάνεν από την Κομισιόν. Um, Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, κύριοι βουλευτέ, με χαρά θα σα παρουσιάσω την απόφαση που υιοθετήθηκε στι αρχέ του έτου, έτου στο Γενάρη και που ακολουθήθηκε από διάφορα μέτρα συνοδευτικά, κάποια από τα οποία αναφέρθηκαν από διάφορα μέλη εδώ της Επιτροπής. Η αναθεώρηση της, της πολιτικής αλληλείας υποβλήθηκε τον Ιούλιο και προβλέπεται η έγκριση του συνολικού πακέτου τον Νοέμβριο. Έχουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 που επικεντρώνεται στην βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως ξέρετε έχουμε πέντε στόχους που αφορούν την απασχόληση, περιβάλλον, πόρους, εκπαίδευση, μείωση δηλαδή των μαθητών που αποχωρούν από τα σχολεία πρώιμα. Όλα αυτά έχουν ε, γίνει στόχος 7 πρωτοβουλειών που επικεντρώνονται σε αυτά τα θέματα και βεβαίως στην περίπτωση της αλληλείας επικεντρωνόμαστε στους αλληλευτικούς πόρους όπως είπε προηγουμένως η κυρία Βουλευτή. Έχουμε διάφορε επιπτώσει εδώ βεβαίω για την αλία, για το περιβάλλον γενικότερα, αλλά έχουμε και οικονομικέ επιπτώσει όσον αφορά την βιώσιμη αλία, σε σχέση δηλαδή με την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να απολάβουν και αυτέ τι αλληλεία. Αυτές οι πρωτοβουλίες βεβαίως έχουν μακρόπνοο χαρακτήρα. Κάποιες από αυτές έχουν έρθει κοντά στο όριο εκπνοής τους και βέβαια σήμερα θα πρέπει να δούμε πώς θα ισορροπήσουμε τις προσπάθειες οικονομικής βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά το οποίο είναι απαραίτητο. Επίσης, οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ένα ευρύ χαρακτήρα, δηλαδή ασχολούνται και περιλαμβάνουν διάφορους τομείς πολιτικής όπως κλίμα, μεταφορές, ενέργεια, φυσικούς πόρους, πρώτες ύλες, μέταλλα, εδώ έχουμε να κάνουμε με την γεωργία, με την ε, αλία βεβαίως όσον αφορά το περιβάλλον της ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν το σημείο κλειδί είναι το να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε και να συμβάσουμε διάφορους στόχους ώστε να δώσουμε μια οικονομική όθηση ώστε να υπάρχει ανάπτυξη και απασχόληση αλλά ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη χρήση των πόρων και θα πρέπει επίσης να εντοπίσουμε διάφορες νέες ευκαιρίες ώστε να υπάρχει καινοτόμος ανάπτυξη η οποία θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα. Και όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να τεθούν υπό το φως της ε, κλιματολογικής περιβαλλοντικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουμε την επάρκειά μας και την βεβαίως επιβίωση συγκεκριμένων ειδών. Αυτό που προτείνεται είναι ένα συνολικό πακέτο μέσο και μακροπρόθεσμων μέτρων. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο την προοπτική 2020, αλλά έχουμε και συγκεκριμένες δράσεις καθοριστικές, ώστε να φτάσουμε στο 2050 σε περίπου 40 χρόνια, δηλαδή σε μια γενιά και βάλε, αλλά τα βήματα που θα γίνουν σήμερα θα έχουν αντικτύπο σε 40 χρόνια. Αν δείτε πριν 40 χρόνια τι γινόταν στη δεκαετία του 70, πολλά ακόμα ισχύουν από τη δεκαετία του 70, οπότε είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις ανάγκες των μελλοντικών δεκαετιών στις σημερινές μας δράσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία βεβαίως απαιτεί και μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά τις διάφορες συνέργειες και συνεργασίες. Χρειαζόμαστε επίσης άμεση δράση ώστε να εξετάσουν μακροπρόθεσμα τις δράσεις τους οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται σήμερα σε αυτές τις δράσεις από το 2020 δηλαδή, και πέρα μέχρι το 2050. Μία άλλη πτυχή που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Καταναλωτές είναι μία από τις πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις όσον αφορά την παραγωγή. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι και θα πρέπει η καινοτομία βεβαίω να κατευθύνεται στη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίω η Ευρώπη δεν είναι μόνη τη στον κόσμο. Η πολυεθνικές είναι ένα άλλο σημείο κλειδί και στον τομέα της αλληλείας και του χρόνου θα έχουμε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη στο Ρίο, Ρίο συν 20, που θα αφαιρωθεί στην βιώσιμη ανάπτυξη, στη διακυβέρνηση και στην χρήση των πόρων. Και υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη σε συνεργασία με άλλου εταίρου μα στον κόσμο ώστε να καθορίσουμε σωστά τι προτεραιότητε μα Και βέβαια υπάρχουν και διάφορα εργαλεία πολιτική τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα, ώστε να καθορίσουμε προδιαγραφέ, αλλά επίση και εργαλεία αγορά, ώστε να υπάρχουν οι σωστέ τιμέ στην αγορά. Ένα άλλο σημείο κλειδί αυτό. Ένα άλλο σημαντικό επίση είναι η ενημέρωση του καταναλωτή, ώστε ο καταναλωτή να μην βασίζεται μόνο σε γραπτέ πληροφορίε, οι οποίε είναι αρκετά περίπλοκες, αλλά οι τιμές θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες προς τους ε, καταναλωτές για να βλέπουν αν μπορούν να καταναλώσουν κάτι, να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να το καταναλώσουν οικονομικά ή όχι. Η πληροφορία λοιπόν είναι πολύ σημαντική εδώ. Όσον αφορά τώρα την ζήτηση και την προσφορά, και εδώ ε, θα πρέπει να έχουμε μια οργανωμένη συντεταγμένη ε, δράση, όχι μόνο αποσπασματικά, και θα πρέπει βεβαίω να πούμε ότι και η έρευνα και η ανάπτυξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, οπότε θα πρέπει να έχουμε σημαντικές αποτιμήσει αντικτύπου. Γιατί καμιά φορά τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι τα οριστικά. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση από την Κομισιόν, κάτι το οποίο ήδη κάνουμε τα τελευταία τρία χρόνια, για πλήρη και διεξοδικά στοιχεία όσον αφορά τους αντικτύπους, ώστε να τα χρησιμοποιούμε αυτά σωστά στη χάραξη των πολιτικών. Νομίζω ότι ο στόχος οποιασδήποτε πολιτικής είναι το να έχουμε κατάλληλους στόχους και πολιτικές και να δούμε ακριβώς πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά με τον καλύτερο, με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για την κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς όπως σας έλεγα χρειαζόμαστε συνεχείς αξιολογήσεις όσον αφορά τον κύκλο ζωής και τα δομένα που τους συνοδεύουν. Θα πρέπει να κοιτάμε δηλαδή τι γίνεται από την αρχή με μετρήσεις, με δείκτες για τους οποίους χρειαζόμαστε εναρμονισμένους δείκτες και στοιχεία και θα πρέπει να έχουμε πλήρη και ενημερωμένα στοιχεία. Οι διάφορες πρωτοβουλίες που προβλέπονται υπό τις πρωτοβουλίες αυτές εν μέρει υιοθετήθηκαν φέτος. Έχουμε τέσσερις μακροχρόνιες ή μακρόπνοες προτάσεις για την οικονομία χαμηλού άνθρακα, για το μέλλον και το ρόλο των ε, μεταφορών, όπως επίσης και για την αλία στην Ευρώπη. Εδώ κοιτάζουμε και άλλα θέματα, άλλους πόρους δηλαδή εκτός από την ενέργεια και τις μεταφορές και νομίζω ότι αυτά τα τρία στοιχεία ήδη οθετήθηκαν στις αρχές του έτους. Έχουμε το τέταρτο που αφορά την ενέργεια που θα υιοθετηθεί τον Δεκέμβριο, δηλαδή έναν χάρτη οδικό για την ενέργεια μέχρι το 2050. Στοιχείο αυτό πάρα πολύ σημαντικό βεβαίω για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που αναφέραμε. Εκτός από αυτή την μακροχρόνια δράση. Έχουμε και συγκεκριμένε δράσει για την ενέργεια, για την αλληλεία και για άλλου τομεί μετά από συγκεκριμένε προτάσει που υπέβαλε η Κομισιόν τον ε, Ιούνιο. Είχαμε κάποιε προτάσει και σχέδια δράση για την βεπικιλότητα μέχρι το 2020 και βεβαίως είχαμε και την αναθεώρηση της ε, αληφθικής πολιτικής που υποβλήθηκε τον Ιούλιο. Είχαμε την ε, Γεωργία επίση και τη μεταρρύθμιση τη Γεωργία η οποία θα υποβληθεί αύριο και είχαμε επίση και την περιφερειακή ανάπτυξη, θέμα το οποίο μα απασχόλησε πρόσφατα. Έχουμε και άλλε προτάσει οι οποίε θα υποβληθούν προ τα τέλη του έτου αλλά και στι αρχέ του επόμενου έτου όσον αφορά την ανακύκλωση, την ε, κατανάλωση, την ποιότητα αέρα και ύδατο. Όλα αυτά έρχονται μέσα στο 2012. Το ορίο συν 20, όπως έλεγα, η διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει μια πραγματική ευκαιρία αλλά βεβαίως ε, δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχουν ε, διμερείς επαφές και διμερείς συνεργασίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διεθνείς εταίροι να συμμερίζονται τις αναλύσεις αλλά και να αποδέχονται την ανάγκη δράσης. Δεν γίνεται μόνο να δρά και να αντιδρά η Ευρώπη και κάποιε άλλε αναπτυγμένε χώρε, θα πρέπει όλοι να δουν ότι υπάρχει ανάγκη για την επίτευξη αυτών των στόχων που ανέφερα και με τρόπο βεβαίω αποδεκτό για όλου. Η διεθνή λοιπόν συνεργασία βεβαίω θα οδηγήσει στην ανταλλαγή δεξιοτήτων και βελτίστων πρακτικών. Επίση, η παγκόσμια ζήτηση αποτελεί μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει που έχουμε μπροστά μα, γιατί τα το επίπεδο ζωής θα αυξηθεί, οπότε αυτό θα συνοδευτεί βεβαίως από αύξηση κατανάλωση η οποία θα εμπνέεται από τον δικό τρόπο ζωής. Αυτό βεβαίως εν μέρη είναι θεμητό, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι τα σφάλματα που είχαμε στις δυτικές και στις αναπτυγμένες χώρες δεν θα επαναληφθούν από τις αναπτυγμένες χώρες, κάτι το οποίο νομίζω το έχουν καταλάβει, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς θα το πετύχουμε αυτό και πώ θα βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Σε σχέση τώρα με τη διακυβέρνηση και την ε, επιτήρηση και την παρακολούθηση της πρόοδου, νομίζω ότι όλος ο στόχος της στρατηγικής 2020 βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη. Και αν τα κοιτάξουμε όλα αυτά σε σχέση με την προηγούμενη στρατηγική της Λισαβόνας, βλέπουμε ότι έχουμε ένα ευρύτερο μεγαλύτερο οριζόντα μέχρι το 2050 και ακόμα παραπέρα ενδεχομένω. Η Ευρώπη λοιπόν 2020 περιλαμβάνει δράσει μέσω και μακροπρόθεσμες, οπότε κατά την άποψη της Κομισιόν θα ήταν σημαντικό να ενσωματωθούν και οι δύο αυτές στρατηγικές σε μια διαδικασία διακυβέρνησης, ώστε να βρούμε τις καλύτερε δυνατέ συνεργασίε, ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσει και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου θα μπορούσαμε να δούμε το όλο θέμα σφαιρικά. Αυτό που νομίζω είναι απόλυτα απαραίτητο είναι οι πληροφορίε να υποβάλλονται με τρόπο εύπεπτο, δηλαδή οι δείκτε για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να είναι αρκετά λειτουργική ώστε να βοηθούν ακριβώ τη χάραξη τη πολιτική. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε είναι το να χτίσουμε σε αυτά που ήδη έχουμε διαθέσιμα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε επίση ότι Πρέπει να εντοπίσουμε τα κύρια στοιχεία, τα οποία ενδεχομένω θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε στοιχεία πολιτική και που θα μα βοηθήσουν στη χάραξή του. Και όπω είπα συγκεκριμένα, η Κομισιόν έχει υποβάλει προτάσει για διάφορου ε, τομεί. Βεβαίω, σα αφορά εδώ το θέμα τη αλληλεία. ως ε, κοινοβούλιο βεβαίω ακόμα περισσότερο και έχουμε καλέσει όλου του εμπλεκόμενου να συμμετάσχουν, να υποβάλουν τι προτάσει του. και να το κάνουν μέσω συζητήσεων οι οποίες θα αφορούν συγκεκριμένε προτάσεις. Ο πρόεδρος Κομισιόν νομίζω υπό τη δική του ευθύνη για να υπογραμμίσει την ε, πολιτική σημασία διατύπωσε αυτέ τι πρωτοβουλίε, αλλά τσάφησε ακριβώ και ενέ περιεχομένου ώστε να συμπληρωθούν από τι προτάσει των ε, διαφορών εταίρων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία τρότμα για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ την Κομισιόν επί ευκαιρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμήσαμε σίγουρα στο ότι είμαστε σε θέση ε, να δούμε σε ευρία γωνία, θα λέγαμε, ευρέως την πολιτική την Επιτροπή. Θα ήθελα όμως η παρουσίαση που έγινε σήμερα το πρωί από την Επιτροπή να είναι πολύ πιο επικεντρωμένη. Ε, διότι ασχολούμαστε με την μεταρρύθμιση της κοινή ελληνική ε, πολιτικής και αυτό που θέλουμε είναι να συμβάλλουμε ε, πάνω σε προτάσεις συγκεκριμένες, διότι οι αλληλείς και όλος αυτός ευρέως ο επαγγελματικός χώρος περιμένουν από εμά να σκύψουμε πάνω από τα πρόβλημα τους και ενδιαφέρονται ε, τόσο για την προστασία των πόρων όσο και την ανάπτυξη αυτού του χώρου. Πάνω σε αυτά εμείς θα επιμείνουμε Πρέπει να δούμε τις οικονομικές πτυχές ε, και γι' αυτό το θέμα θα θέλαμε να κάνουμε μια έκκληση άλλη μια φορά προς την Επιτροπή να δει το θέμα αυτό και όσον αφορά την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την οικονομική διάσταση όσον αφορά ε, την ανάπτυξη του αλλιευτικού τομέα στην Ευρώπη. Αυτά σε σχέση με την παρουσίαση που μας έγινε από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Τρότμαν. Ελπίζουμε στην επόμενη συνεδρίαση να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάντως την Κομισιόν. Θα πέρασουμε στο σημείο 10. Μελέτη για τις προοπτικές του Νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Όπως ξέρετε, αποφασίσαμε να ζητήσουμε τη διεξαγωγή μια μελέτη για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία. Οι προτάσει δεν έχουν υποβληθεί ακόμα από τον Αρμόδια Επίτροπο και πριν από λίγου μήνε η υπηρεσία μελετών έχει υποβάλει μία μελέτη την οποία θα έχετε ήδη δει και επί τη ευκαιρία να καλωσορίσω την κυρία Ιντράνη Λούτσμαν και την κυρία Σοφή Ντεκλέρ εμπειρογνώμονες για τα θέματα αλληλείας είναι εδώ νομίζω τις καλωσορίζω και θα δώσω το λόγο καταρχήν στην κυρία Λούτσμαν να μας κάνει μια παρουσίαση 20 λεπτά το πολύ. Έχετε το λόγο κυρία Λούτσμαν. Thank you, Madam Chair. Um, as, as someone Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, η κοινωνική πολιτική βρίσκεται υπό αναθεώρηση και αναλάβαμε λοιπόν την εκπόνηση αυτής της μελέτης με δύο στόχους. Για καταρχήν να εντοπίσουμε και τις κύριες οικονομικές ανάγκες του τομέα αφενός και να αφετέρου προτείνουμε τρόπους για την μελλοντική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ελίας. Θα αναφερθώ σύντομα στην ανάλυση που κάναμε και μετά θα αναφερθώ σε κάποια άλλα σημεία στην παρουσίαση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πω σύντομα τα εξής. Η μελέτη αυτή που κάναμε ήταν σύντομη. Αναθεωρήσαμε και εξετάσαμε όλα τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Αλληλευτικό Ταμείο και κάναμε και μία έρευνα online Στη συνέχεια κινητοποιήσαμε εμπειρογνώμονες για θέματα προπολογισμού και κάναμε κάποιο brainstorming για τα πιθανά μελλοντικά σενάρια. Τώρα, η αξιολόγησή μας για αυτό το ταμείο έχει διάφορα αποτελέσματα. Το πρώτο είναι ότι κοιτάξαμε το πώς γίνεται ο προγραμματισμός για το αλευτικό ταμείο. Και η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά, γιατί στην ουσία το ταμείο αυτό αποτελεί μια συνέχεια του FIG Παρ' όλα αυτά οι δράσεις και τα μέτρα είναι αντικείμενο διαφορετικής οργάνωσης. Ο προγραμματισμός είναι ένας άλλος μηχανισμός και πολύ συχνά τα μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άλλο εθνικό πρόγραμμα και άλλο στρατηγικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο επιφέρει μεγάλο φόρτο Δουλειά όσον αφορά το Ταμείο Αλίας. Παρ' όλα αυτά, οι μηχανισμοί, παρόλο που ήταν αρκετά δυσκίνητοι, δεν επέτρεπαν στο να αναπτύξουμε την εταιρική μας σχέση με τους εμπλεκόμενους. Και εμείς αναγνωρίζουμε ότι αυτό ακριβώς αποτελεί και τη μεγάλη διαφορά για το πρόγραμμα για το αλληλευτικό ταμείο. Δηλαδή για πρώτη φορά συμμετείχαν οι εποφελούμενοι, οι συμμετέχοντες από την αρχή, από τη χάραξη του, του προγράμματος. Το 2008 είχαμε ένα επιπλέον σημείο το οποίο προσθέθηκε στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας, το οποίο, να το πω έτσι απαλά, δεν βοήθησε και πάρα πολύ τον προγραμματισμό γιατί επέφερε περισσότερη εργασία και αυτό ακριβώς ήταν το αντικείμενο μιας εκ των συστάσεών μας. Ότι δηλαδή θα πρέπει τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ξεκινάνε από την αρχή και να μην συζητιούνται όσο προχωράει η εργασία αυτή. Και τέλος, το EFF περισσότερο από το EFIG χρειάζεται ένα περισσότερο ολοκληρωμένο έλεγχο και διαχείριση σε βαθμό μεγαλύτερο, θα έλεγα, από ότι πριν. Βεβαίως αυτό σημαίνει θα πρέπει να δημιουργούνται καθυστερήσεις, αλλά θα πρέπει αντίθετα να έχουμε το κατάλληλο εργαλείο στην ε, διάθεσή μας το οποίο θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι νέε ε, διατάξεις όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και κυρίως τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης προκάλεσαν πάρα πολλές καθυστερήσεις στην εφαρμογή και η προγραμματική περίοδος ξεκίνησε το 2007 ή θα έπρεπε να ξεκίνησε το 2007 και όπως θα δείτε από τα στοιχεία εδώ για κάποιους δεν ξεκίνησε παρά το 2011 και μόνο αφού ε, επικυρώθηκε το IMCS. Οπότε η ερμηνεία μας εδώ είναι ότι όντως υπήρξαν καθυστερήσεις από την αρχή, αλλά τα προβλήματα της Κομισιόν αφορούσαν την καθυστερημένη οθέτηση των κανονισμών, την καθυστερημένη έκδοση κατευθυντήριων γραμμών, οπότε όλα αυτά προκάλεσαν καθυστερήσεις. Και δεν είχαμε μόνο να κάνουμε με τις νέες χώρες μέλη, Όλες οι χώρες νομίζω αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω ακριβώς της αντίθεσης μεταξύ του εθνικού και του υποεθνικού, περιφερειακού δηλαδή επίπεδου. Τώρα για τις τρέχουσες ανάγκες. Και το συμπέρασμά μας ήταν ότι αυτή η εταιρική σχέση με τους εμπλεκόμενους τι σήμαινε, ότι τα εθνικά προγράμματα αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ανάγκες του κλάδου και χρειάζεται να υπάρχει καλή στρατηγικός προγραμματισμό, διότι είπαμε ότι αυτές οι τρέχουσες ανάγκες του κλάδου, όπως τι αποτυπώνει η η πράσινη βίβλος και όσον αφορά αυτή την εκ αξιολόγηση του FIFG καλύπτονται. Και είπαμε ότι καλύπτονται αυτή εξ αρχής αυτή η συμμετοχή και παρόλα αυτά το, το, πρόγραμμα ε, δεν έχει λογική παρεμβατική όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο και όσον αφορά την παρέμβαση οργανωθήκαμε με τέτοιο τρόπο που καθίσταται αρκετά δύσκολο τόσο ώστε να μπορούμε να δούμε τους ε, ε, δείκτες, τους μακροοικονομικούς ή τέλος πάντων τους μακροδείκτες και είπαμε ότι δεν υπάρχει σύστημα πληροφορικής που να δίνει δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο στην Κομισιόν ε, να, να μπορέσει να ελέγξει με κάποιους ε, αιτήσους δείκτες το πώς τα κράτη-μέλη αξιοποιούν τα κονδύλια. Ούτε υπήρχε κάποιο είδους ε, δείκτης για τις ε, επιπτώσεις στην αρχή. Επομένως, το ότι ξεκινήσαμε καθυστερημένα σημαίνει ότι ε, η εφαρμογή ε, ήταν πάρα πολύ πρόημη διότι μόνο το 15% του προπολογισμού του EFF ε, είχε εκταμιευθεί και η ενδιάμεση αξιολόγηση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα flags του Farnet ήταν τη μόνη θετική επίπτωση του τέταρτου άξονα. Τώρα, μέλουσες ανάγκες του κλάδου. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερη απόδοση του EFF. Και η σχετική έρευνα των εμπλεκομένων μας έδειξε ότι υπήρχε περιορισμένη εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος. Και αυτό γιατί είχαμε χρηματοδότηση και από τους δικαιούχους και από το κράτος. Άρα θα πρέπει στο μέλλον να υπάρχει αρρωγή από την Κομισιόν που να είναι έγκαιρη και φιλική στο χρήστη να υπάρχει περισσότερη λογική πανεμβατισμού στο πρόγραμμα. Βλέπετε τώρα εδώ, α, μία διαφάνεια την ε, παραλείψαμε, ίσως επανέθουμε, αλλά θέλω τώρα να σας δείξω ποια είναι η λογική του προγράμματος του EFF και μπορεί να δείτε εδώ με αυτές τις αξιολογήσεις ε, και βλέπετε ε, τα, τα μέτρα αυτά τα οποία είναι μέσα στα κουτάκια πώς ε, συνδυάζονται με αυτήν την παρεμβατική λογική. Ναι. Uh, with the recommendations from the first task. Um, she highlighted three important areas. Ναι, θα σας αναφέρω τρεις σημαντικούς τομείς δράσεις για το μέλλον. Να πω όμως ότι κατάξαμε στο συμπέρασμα ότι το μελλοντικό θαμείο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πολιτικές βιώσιμης. Διαχείριση σπόρων. Έχουμε και την πολιτή, το πολιτές πλαίσιο που θα καλύψει το 2014 μέχρι το 2020 με κάποιες πολύ σημαντικέ αλλαγές οι οποίε θα έχουν επίπτωση στον τομέα. Θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Προσπάσαμε λοιπόν να εστιάσουμε σε όλα τα παραπάνω στοιχεία και να κάνουμε τι απαραίτητε αναλύσει, να δούμε επίση τι μελλοντικέ εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε ακριβώ πώ θα μπορούσαμε να τα εσωματώσουμε όλα αυτά στο μελλοντικό EFF. Αν δείτε εδώ αυτά που λέει η διαφάνεια, αυτό που κάναμε και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο ένταξη των βημάτων τη μελέτη αντικτύπου όπου καταρχήν έχουμε τους στόχους οι οποίοι καθορίζονται. Και είδαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να εντάξουμε αυτά τα αποτελέσματα των μελετών στο μελλοντικό πρόγραμμα είναι να βρούμε κάποια σενάρια, κάποιες ε, εναλλακτικές λύσεις και εμείς κάτσαμε εδώ και επεξεργαστούμε τέσσερις, 0, 1, 2 και 3. Και το EFF παραμένει ε, το κλειδί για αυτή την ε, πολιτική στην εναλλακτική 0 ε, το EFF ε, παραμένει αμετάβλητο με στόχους, άξονες και μέτρα που έχουν τη σημερινή μορφή αλλά και περιεχόμενο. Ε, δεύτερη επιλογή, παίρνουμε λαμβάνουμε υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης και γιατί είπαμε ότι εδώ δεν υπάρχει ισχυρή πανεμβατική λογική και όπως είπαμε ε, θα έχουμε τροποποίηση στην αρχιτεκτονική του. Αλλά όμω ο πυρήνα, η ιδέα κεντρική παραμένει ουσιαστικά ίδια. Στη δε, δεύτερη επιλογή, την υπαριθμών 2, πάμε λίγο παραπέρα και λαμβάνουμε υπόψη κάποιες εξελίξεις ε, που αφορούν το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο στον προπολογισμό της Ένωσης και λέμε ότι θα πρέπει η αρχιτεκτονική να ε, είναι όπως πριν αλλά αλλάζει ο πυρήνας, η καρδιά του προγράμματος και θα πρέπει να υπάρχει βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων. Και υπάρχει μια άλλη επιλογή, η υπαριθμόν 3, αφορά ε, το ότι ε, το Ταμείο τώρα θα υποστηρίζει τις παράκτιες κοινότητες. θεωρείται αυτή κάπως πιο ακραία η επιλογή. Η διάκριση επίσης μεταξύ του status quo και της πρώτης επιλογής και μια άλλη μεριά της δεύτερης και τρίτης είναι το ότι θα πρέπει να μην είναι ακατανόητα τα μέτρα και να βλέπουμε οι αυτοί οι άξονες κατά πόσον θα παραμείνουν θα καταργηθούν. Στο status quo και σε αυτό που λέμε επίσης οψιόν πρώτη, επιλογή πρώτη, εξαρτάται πολύ από τα κράτη-μέλη για τις επενδύσεις. Τα 2 και το 3 όμως θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους μεταβατική διαχείριση με καινούρια μέσα πολιτικής σε επίπεδο κοινοτήτων. Τώρα, εάν έχετε το κείμενο μπροστά σας, πηγαίνετε στο 14-15 από τις διαφάνειες για να δούμε αυτά τα οποία ξεκίνησαν από την Πράσινη Βίβλο σαν ερωτήματα. Αφού επεξεργαστήκαμε αυτές τις επιλογές, αυτά τα σενάρια, θέλουμε να δούμε η καθεμία από αυτές πώς καλύπτει τα ερωτήματα που τίθενται στην Πράσινη Βίβλο. Η επόμενη διαφάνεια τώρα. Α, δεν μπορεί να τη δείτε αν κάθεστε πίσω, είναι πολύ μικρά τα γράμματα, αλλά Θέλω να δούμε δύο σημεία εκεί που λέει η option 1. Πώς καλύπτει τα ερωτήματα της πράσινης βίβλου για, για τον άξονα Y και μετά λέει τον άξονα Χ. Βλέπετε τρόπο πώς αλλάζει η αρχιτεκτονική του ΙΒΕΦ στο μέλλον και πώς ε, αρχίζει η παρεμβατική λογική να μπαίνει περισσότερο. Μπορείτε επίσης να δείτε εδώ πέρα ότι εδώ ε, μπαίνει το θέμα του, της μεταβατικής διαχείρισης και, και να υπάρχει μεριωτός συντονισμό, όχι μόνο με την πολιτική της θάλασσας αλλά και με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή αλληλευτική πολιτική και είδαμε πώς θα λάβει μεγάλες τις διαστάσεις ε, η αλληλεία μικρής κλίμακας. Μετά πάμε στην οψιόν 2. Και για να δούμε τι κάνει αυτή, τι λέει αυτή για τα ερωτήματα της Πράσινης Βίβλου, αν διοργάνωσε του ΕΦΕΦ, e κατάργησε το άξονα 1, μπορείτε να διαπιστώσετε εδώ, αλλαγή, ε, σε, οι πόροι να πηγαίνουν σε καινοτομία, νέα μέσα πολιτικής, νέα εργαλεία πολιτικής, ισότητα μεταχείρισης για όλο τον, τον κλάδο, ιδίως όσον αφορά την αλία μικρής κλίμακας. Αν διαβάσετε τι να σας πω, 20 λεπτά τι, πού να τα καλύψω αυτά. We went to that point of, of how well does our options... Uh, για να δούμε λοιπόν αυτές οι λαϊκές λύσεις πόσο καλά απαντούν στα ερωτήματα της φάσης βίβλου. Το 1 και το 2 τα σενάρια λένε για αυτό το ταμείο. Τώρα στο 2 είπαμε πρέπει να αξιολογήσουμε αυτά τις οψιών, αυτά τα σενάρια με κάποιους δείκτες, όχι οικονομικούς αλλά περιβαλλοντικοί δείκτες, κοινωνικοί δείκτες. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά στον πίνακα 12 στην έκθεση. Να και τα συμπεράσματα. Παρακάτω. Σενάριο 1. Αξιολογείται με αυτούς τους δείκτες. Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση. Α, όχι, όχι, για ποιον, μηδέν, μηδέν λέει, μηδέν. Το status quo θα επιδεινωθούν τα πράγματα λόγω των αποθεμάτων, λόγω της κρίσης. Το σενάριο παριθμών 1. Έχουμε την τροποποιημένη δομή του ΙΕΦΕΦ και αναδιοργάνωση στόχων κλπ. Εδώ θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή του ΙΕΦΕΦ. και θα έχουμε κάποιο, κάποιες επιπτώσεις κοινωνικές, περιβαλλοντικές κλπ. Οπότε είπαμε παρακάτω ότι θα έχουμε στην οψιόν 3 κάποια ωφέλεια όσον αφορά ε, την αλία και για την ε, στρατηγική του 2020 θα έχουμε ε, θετικές επιπτώσεις ε, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όμως επίσης πρόκειται να έχουμε αρνητική και ε, κοινωνικές ε, ε, μέσω πρόθεσμα. Και οπότε θα πρέπει να περάσουμε από μία μεταβατική περίοδο για ένα νέο ταμείο ελίας όπου θα έχουν αλλάξει πάρα πολύ βασικές παράμετροι. Η τελική, η τελευταία τώρα, ο, ο τελευταίο ε, σενάριο λέει ότι θα υπάρξουν ωφέλειες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές και επίσης θα βοηθηθούν με, βιώσιμο τρόπο οι παράκτιες αλληλευτικές κοινότητες. Συμπεράσματα τώρα. το σενάριο 0. Ε, εδώ είναι το status quo. Όπως είπαμε, είπαμε ότι δεν είναι βιώσιμο σενάριο όπως έχει σήμερα η συγκυρία. Και επίση, όσον έχουμε την κρίση, έχουμε την κατάσταση των αποθεμάτων, η προβληματική συνεχίζεται και μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχει οικονομική κρίση σε όλα τα κρατημέρια και επομένως δεν είναι βιώσιμο αυτό το σενάριο το, το 0. Ε, ε, σενάριο 1 λέμε ότι θα πρέπει να δούμε πόσο χρειάζεται μια μεταρρύθμιση στο EFF αλλά δεν δείχνει αυτό το σενάριο ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν σε σχέση με την δέουσα μεταρρύθμιση. Πάρα assets um, do most in the transition to a resource efficient. Θέλουμε εδώ πέρα παρακάτω να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδους πιο αποτελεσματική οικονομία, ε, πιο αφιλική στο περιβάλλον, δεν ξέρω πώς θα τα δείτε, αλλά το δικό μας συμπέρασμα είναι ότι το δεύτερο σενάριο είναι το πιο ρεαλιστικό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, το D3 είναι πιο, πιο, πιο ριζοσπαστική αντίληψη για αυτό το Ταμείο της Αλίας. Ε, πιο δύσκολο να περάσει. Um, I'm sorry if we ran over time, um, but hopefully we'll uh, be able to entertain some questions from the committee. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις που έχει η Επιτροπή. Eh, eh, Πρόεδρος, κοιτάξτε. Σας ευχαριστούμε. Εγώ διάβασα όλο σας το κείμενο. Και η κυρία Λέβιν έχει ζητήσει το λόγο. Thank you very much and thank you for the... Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και για την εισήγηση. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση του υπάρχοντος EFF. Μας είπατε ότι τα κράτη-μέλη όσον αφορά την οικονομική βοήθεια ε, αυτή η βοήθεια αντιστοιχεί σε μία συρρήγνωση του στόλου περίπου κατά το ίμιση. Έχουμε το θέμα της οικονομικής κρίσης, τη σύγκνωση των ε, πόρων, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να δούμε ποια είναι η επίπτωση της κρατικής παρέμβασης για τα αποθέματα. Άρα συστήλετε για τις ενισχύσεις. Αυτές οι, οι ενισχύσεις τύπου scrap βοήθησαν ου. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Well, Α, πολύ δύσκολο το ερώτημα, λέει ο Μιλήτρια. Όχι, όχι, δεν σας πω την προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω ότι από τα στοιχεία που έχουμε, σίγουρα δεν είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε αν αυτές οι επιδοτήσεις στα πλαίσια του ΕΦΕ θα έχουν βοηθήσει όχι, αλλά από την αξιολόγηση του προηγουμένου καθεστώτος για το EFF καταλήξαμε στο ότι περιπτωσιολογικά μόνο κανείς μπορεί να καταλήξει εάν έχουν κάνει τη διαφορά όταν υπάρχουν κοινά αποθέματα για στα κράτη-μέλη, όταν υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες ε, λειτουργίες των εμπλεκομένων, δεν βγαίνει άκρη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε ακόμα να καταλήξουμε ε, κάπου για αυτές τις επιδοτήσεις. Γκάλαχερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βλέπω σε αυτή τη συνοψή ότι μόνο 15% του προπολογισμού ήταν ενισχύσει το 2010 και εκταμιεύτηκαν. Και λέει εδώ πέρα είναι πολύ νωρί να... Τι λέει η Κομισιόν. Πολύ νωρί λέει για την αξιολόγηση. Τι θα κάνουμε. Θα εκταμιευθούν αργότερα τα χρήματα ή όχι. Αν ε, δούμε την κοινή γεωργική πολιτική θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει πρόγραμμα ανάπτυξη Πέτρο που έχει βοηθήσει και για ένα μελλοντικό αλληλευτικό ταμείο, ταμείο για την αλληλεία τέλο πάντων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολιτική για την υπεθρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά αλληλευτικά λιμάνια που έχουν απεριμωθεί και εκεί θα έπιαναν τόπο τα κοινωνικά χρήματα. Θα δίναμε πνοή ζωής. Όχι αναγκαστικά να ασχοληθούμε με την αλληλεία, όπως να ενισχυθούν ο του τουρισμού, να φτιάχνουμε καμιά μαρίνα. Να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Εγώ απλά ήθελα να το επισημάνω τώρα, Πρόεδρε. Είναι παλιό το πρόβλημα. Είπαμε, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στην ΚΑΠ. Έχουμε καθήκον προς αυτές τις κοινότητες. Δεν φταίνε εκείνοι που έχουν συρρυκνωθεί τόσο πολύ τα αποθέματα, οι εκφορτώσεις αλλιέων κλπ. Οπότε θα μπορούσαμε να τους δώσουμε μια τέτοια όθηση να πάνε προς τα μπρος. Just to also continue the discussion that Mr. Αρσένης. Γι' αυτό είπα και κ. Γκάλαχερ. Με το Γεωργικό Ταμείο υπάρχει χρηματοδότηση. Αν θέλουμε να τα κάνουμε αυτά τα λιμάνια τόπους τουρισμού. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει το Ταμείο να χρησιμοποιηθεί για να σώσουμε ψάρια και ψαράδες. Όταν ξεκίνησε η αληθική πολιτική, αυτό που θέλαμε είναι να πετύχουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και επενδύσαμε σε αυτό. Τώρα. Τα ψάρια τώρα τόσο λίγα που δεν μπορούμε ούτε καν να τα βρούμε, να ασχοληθούμε με την κοινή πολιτική σε μερικά μέρη. Αλλά θα πρέπει να ασκήσουμε κάποια πολιτική. Και φυσικά θα πρέπει να πάνε χρήματα σε, αυτές, σε αυτά τα μικρά λιμάνια αλλά θα πρέπει να συνδεθούν με, με αλία αυτά τα κονδύλια και να λάβουμε υπόψη το πώς θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους όσον αφορά τα αποθέματα. Γιατί υπάρχουν ε, ληφτικοί πόροι, υπάρχουν ψάρια. Και άρα μπορεί να υπάρχει δραστηριότητα. Yeah, Λέβιν. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό που ρώτησα για τις επιδοτήσεις σκραπ. Πώς θα αποκτήσουμε περισσότερες παραγωγικές δυνατότητες, τι θα κάνουν τα κρατημέλη. Κάποια κρατημέλη έχουν πάρα πολύ κακή επίδοση όσον αφορά τα στατιστικά που υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και για την απασχόληση. Τι, τι θα γίνει. Για πέστε μας. Um, yes, actually that, that refers more to another bit of work that IEP did on looking at the capacity of the European fleet. Έχουμε ετήσιες εκθέσεις και από το STCF έχουμε νέους δείκτες που βέβαια δεν μας καλύπτουν, μας λύνουν το πρόβλημα. Αλλά για το ελευτικό ταμείο δεν ήταν δυνατό να γίνει τέτοιο συσχετισμό. Οπότε κάποια λίγα κονδύλια τα οποία θα αφορούσαν τον πρώτο άξονα όντως ήταν από το αληθικό ταμείο. Και έτσι μπορέσαμε να συνδέσουμε τις, τις αληθικές δυνατότητες και την θρησιμότητα των ψαριών με το ταμείο. Άρα, δυστυχώς, προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει και εκείνη το λόγο για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία ερωτήματα υποβλήθηκαν, ευχαρίστως να απαντήσω. Πρώτον. Eh, για τις δημοσιομικές προοπτικές έχουμε να πούμε ότι θα πρέπει να δούμε αν θα καλύψουμε κάποιες τέτοιες κοινότητες. Η απάντηση είναι ναι. Με κάθε επιφύλαξη για το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά το χρηματοδοτικό μέσο που έχουμε ανακοινώσει, καταρχήν αυτή η πρόταση θα εγκριθεί τέλη Νοεμβρίου. Και η Επίτροπος Δαμανάκη ξεκάθαρα έχει δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που με επιφύλαξη της τελικής γνώμης της Επιτροπής θα πάρουν τα πράγματα έτσι στον δρόμο τους. Και βασική κατευθυντήρια γραμμή είναι ότι η Επιτροπή θα ακολουθήσει τον τέταρτο άξονα του Ταμείου. Εκείνο δηλαδή που αφορά την ανάπτυξη και την ε, ε, ποικιλία στις δραστηριότητες των παρακτήων κοινοτήτων. Γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτές τις μικρές παράκτιες κοινότητες που πολλές από αυτές εξαρτώνται οικονομικά από την αλληλεία. Και ποτέ εδώ δεν είναι πια είπαμε θέμα αηλίας αλλά θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ευρύτερα για να βοηθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη αυτών των ζωνών και ας μην αφορούν αγκαστικά την Αλεια. Άρα έτσι θα ενεργήσουμε με βάση αυτόν τον άξονα. Να υπάρχει συμπληρωματικότητα στην οικονομική ανάπτυξη με την αλία. Αλλά πάντοτε να έχουμε κατά νου το πώς θα βοηθήσουμε αυτές τις τοπικές μικρές αλληλευτικές κοινότητες. Άρα, καταφατική είναι η απάντηση σε αυτό το οποίο είπατε είναι στόχος μας. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Άλλος στόχος είναι το να βοηθήσουμε την προσαρμογή της κοινή ελευθερικής πολιτικής με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Άρα, προσαρμογή της αλίας, του στόλου για τις απορρίψεις για τους, για, την, ε, για τους πόρους και για το περιβάλλον. Πώς θα τα προστατεύσουμε. Τέλος, όσον αφορά αυτές τις επιδοτήσεις και, την, και τον στόλο και σε αυτό έχει τοποθετηθεί η Επιτρόπος Δαμανάγια. Η πρόταση της Επιτροπής θα επηρεαστεί από μία μελέτη που τώρα ολοκληρώνεται. Μελέτη του ε, Ελεκτικού συνεδρίου. Ε, εκεί αναλύεται το πώς θα γίνει σωστή και επαρκής διαχείριση των πόρων του φορολογουμένου που να πιάνουν τόπο και να μην δίνουν απλώς περιορισμένα αποτελέσματα. Με αυτό ασχολείται τώρα το ελληνικό συνέδριο. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λογικά θέλει να λάβει υπόψη αυτά τα συμπεράσματα της ε, μελέτης αυτής του Κοινωνικού Συνεδρίου. Πρόεδρος. Επιτρέψτε να σας πω το εξή Όσον αφορά την κυρία Δαμανάκη, ήδη αυτό ανεφέρθη. Δεν ξέρω τι θα πει το συνέδριο. Τι να πω. Άλλη παρατήρηση να λέμε ότι η διορθωτική πολιτική και τα προγράμματα των κρατών μελών είναι, ε, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει όσον αφορά τις απορρίψεις. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει αν θα μας οδηγήσει σε προστασία των πόρων. Θα πρέπει να υπάρχει διορθωτική πολιτική που να σε οδηγήσει σε ένα εναλλακτικό μοντέλο προστασίας των πόρων, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Αυτό το οποίο έφταιγε ήταν το πρότυπο που είχαμε, η μέθοδος που είχαμε για την προστασία των πόρων και για τη διαχείριση. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Πρώτα πρώτα είχαμε πει να δούμε τι θα γίνει με τις απορρίψεις. Και μετά έχουμε πάρα πολλά αλληλευτικά σκάφη που είναι πολύ παλιά. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά να μην μειώσουμε την αλληλευτική δυνατότητα. Μην μειώσουμε το στόλο. Και θα πρέπει να αλλάξουμε τη μέθοδό μας, το μοντέλο που ακολουθούμε, γιατί με το παρόν μοντέλο δεν καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και τι έκαμε. Είναι πανάκια το Ταμείο Ηλίας. Δεν νομίζω. Πατράω Νέβες. Επιτρέψτε μου να πανέλθω σε ένα ερώτημα το οποίο δεν και είναι σημαντικό. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελλήνε και ελέγχθη ότι το Ταμείο θα πρέπει να προσαρμιστεί στις νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό ζητώ από την Επιτροπή να μας πει. Λαμβάνει, βάλει υπόψη την προσαρμογή που πρέπει να, ε, να γίνει σε σχέση με τις διάφορες περιφέρειες, τις ειδικές ανάγκες. Έχουμε ακούσει πολλές κριτικές και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασκήσει κριτική εξάλλου για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει η Επιτροπή της προτάσεις όσον αφορά το θέμα των περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις κριτικές που έχουν γίνει, τι ακριβώς γίνεται. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, θα προβλέψει, θα προσαρμοστεί όσον αφορά ε, το θέμα αυτό, τη διάσταση αυτή και με τις απαιτήσει που υπάρχουν σε σχέση με την ε, περιφερειακή διάστασή του. Καλώς λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ναι. Θα το συζητήσουμε αργότερα για αυτό το θέμα. και μιλάμε και πείτε μου τι θέλετε. Ναι, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μόλις είπε η Πρόεδρος. Το θέμα νομίζω, μεταξύ άλλων, είναι το εξή το προηγούμενο ταμείο, νομίζω Αλίας, επιδίνωσε την κατάσταση όσον αφορά τις θάλασσες, τους αλληλείς και τα αλλιεύματα. Και αυτό είναι το θέμα ουσίας νομίζω. Σήμερα η προσέγγιση του νέου ταμείου θα πρέπει να απορρέει από μια διαφορετική πολιτική η οποία θα πρέπει να χαραχτεί. Εξάλλου, εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτή η φυγή προς τα μπροστά. Δηλαδή, σαν να έπρεπε να αποφασίσουμε εκ των προτέρων πώς θα χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο, πριν δηλαδή να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε την μεταρρύθμιση της αλληλείας και του τρόπου διαχείρισή της, διαχείρισης της. Νομίζω ότι η συζήτηση θα πρέπει να ήταν λίγο πιο συγκεκριμένη και θα πρέπει να δούμε καταρχήν τις επιπτώσεις της ανθεώρησης της πολιτικής. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται όμως αργότερα, όχι πριν. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ ανακατεύουμε θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια, οπότε θα κλείσω τη συζήτηση, να ευχαριστήσω τις δύο ομιλήτριες για την παρουσίαση αυτής της μελέτης που θα είναι χρήσιμη για τις περαιτέρω εργασίες μας και νομίζω ότι θα πάμε στο επόμενο σημείο της εμίσιας διάταξης, δηλαδή το πακέτο μεταρρυθμίσεων. En primer lugar está el punto duodécimo, que es la presentación, eh, no, perdón, el punto decimotercero, que es la comunicación sobre la reforma de la política pesquera. 13ο σημείο, ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριος Αλαβράκος. Κύριος Αλαβράκος όμως ε, λείπει σήμερα, οπότε θα ζητήσω εφ' εξής, όλοι οι συγητές για το πακέτο μεταρρυθμίσεων να έρχονται τακτικά εδώ σε αυτές τις συνεδριάσεις. Διαφορετικά η κατάσταση θα είναι χαόδης και θα ήθελα να διατυπώσω ένα παράπονο. Χθε μία από τις συζυγήτριες μας είπε ότι δεν ήξερε ότι είναι συζυγήτρια. Ο κ. Σαλαβράκος σήμερα για την μεταρρύθμιση απουσιάζει. Οπότε νομίζω ότι είναι ελάχιστα σοβαρό το η στάση που έχει αυτή η ομάδα. Τέλο πάντων, πάμε στο σημείο 14. Κοινή ελευθερική πολιτική. Η συγγήτρια κυρία Ρόντουστ. Δεν ξέρω αν καταρχήν θέλει να μιλήσει η κυρία Ρόντουστ, η συγγήτρια, ή να δώσουμε το λόγο πρώτα στην Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, πολύ σύντομα να πω πώς βλέπω τον τρόπο που θα προχωρήσουμε στο χρόνο-διάγραμμα. Όπως και να έχει το θέμα, νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο και οι μεν και οι δε για να σκύψουν πάνω αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε σωστά πάντως προετοιμασμένοι. Τόσο τα μέλη όσο και οι σιώδεις ε, ε θα πρέπει να δουλέψουν καλά, να συνεργαστούν και με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να οργανώσουμε το έργο μας και να διαρθώσουμε καλά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, θα υπάρξει ένα έγγραφο εργασία με το οποίο θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συζητήσεις. Από το 2012 θα το έχετε αυτό το έγγραφο. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας για να γίνει μια σωστή αξιολόγηση τη κοινή αλληλευτική πολιτικής. Δεν θα πρέπει συνεχώ να ξανανοίγουμε το διάλογο, να επαναρχόμαστε. Θα πρέπει να θίξουμε τα σημαντικά και δυνατά σημεία ε, για να τα δούμε στις συνεδριάσεις όπου λαμβάνουμε ε, μέρος. Σκέφτομαι θέμα των, της απορρίψεως των ε, αλλιευμάτων, την, ε, περι, την περιφερειακή διάσταση και ανάλογα θέματα. Θα συζητήσω φυσικά με τον Σιώδη Σίτη, διότι εκτός από την Επιτροπή μας θα πρέπει να έχουμε και ένα ικανό αριθμό ε, Θα πρέπει η Επιτροπή δηλαδή όχι μόνο να κάνει μόνη της τις δικές προτάσεις, αλλά σίγουρα να συζητήσει και μαζί μας ε, κάποια θέματα, εναλλακτικέ λύσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν και να συζητηθούν με το Βαρτακό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, χθε μίλησα με το Σιώδη Ισίτη. 2012 λοιπόν θα έχουμε πολλές ακροασίες, Φλεβάρι, ανταλλαγή απόψεων με προσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το Μάρτι μετά συζήτηση για, την, ε, ε, για το διάσταση που έχει να κάνει με τις περιφέρειες και για να μπορέσουμε να εντάξουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στην έκθεσή μας, θα θέλω η έκθεσή μου να παρουσιαστεί το Μάιο σε μια έκτατη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Ε, η ψηφοφορία 10 Ιουλίου θα μπορεί να γίνει στην Επιτροπή μας και η πρώτη ανάγνωση θα πρέπει να γίνει στην πρώτη ε, Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ λοιπόν για την ε, συμμετοχή όλων σας, συνδρομή όλων σας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, από ό,τι κατάλαβα, θα σας παρουσιάσω την γενική ανακοίνωση σε σχέση με την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος αυτής της πολιτικής. Νομίζω ότι σε αυτό το πακέτο, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο και όπως γνωρίζετε περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, εκ των οποίων πέντε από αυτά εγκρίθηκαν από, την, ε, από το Σύνολο της Επιτροπής τον περασμένο μήνα και ένα από αυτά υπόκειται σε έγκριση η οποία θα γίνει τον Νοέμβριο. Η Κομισιόν λοιπόν θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουμε ως σημαντικό στοιχείο αυτού του πακέτου ένα έγγραφο το οποίο θα προλαμβάνει τρεις βασικούς στόχους. Καταρχήν θα πρέπει να σας δίνει μια εικόνα συνολική για το πώς αλληλοσχετίζονται οι διάφοροι πυλώνες της πολιτικής αυτής. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η πράσινη βίβλος, και ήδη το είπαμε, ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταρρύθμιση της Αλίας είναι ότι υπήρξε ανεπαρκής συνέργεια ή συσχετισμός μεταξύ των διαφόρων πυλώνων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς εφαρμόζονταν με τρόπο κάπως αποσπασματικό σε σχέση με τους άλλους. Για να απλωτήσουμε λοιπόν τη συζήτηση και να είναι η συζήτηση αυτή πλήρης, θα πρέπει καταρχήν να δούμε το εξή. Θα πρέπει να έχουμε ως στόχους, στόχο μάλλον, το να παρουσιάσουμε τα διάφορα στοιχεία τη μεταρρύθμιση και τα νομικά και τα μη νομικά υπό το φως ενό συνολικού πακέτου που θα ήθελε η Κομισιόν να είναι συνεκτικό. Και η συζήτηση αυτή τη ανακοίνωση, η συζήτηση αυτού του κειμένου, θα πρέπει λοιπόν να μα επιτρέπει να υπογραμμίζουμε τις, τους συσχετισμούς, δηλαδή το πώς οι προτάσει αυτού του πακέτου και οι πυλώνες αυτής της πολιτικής σχετίζονται με τους υπόλοιπου. Είναι λοιπόν σημαντικό όταν υποβάλουμε τις προτάσεις να μην περιοριζόμαστε στις ε, νομικές, στα νομικά έγγραφα για τις αγορές, στα νομικά βασικά έγγραφα, στα νομικά έγγραφα για τις οικονομικές ε, προτάσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα συνολικό έγγραφο για το πώς σχετίζονται αυτά και το πώς συνδέονται μεταξύ τους όλα αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό, Πρόεδρε, Όπω ο κ. Βιλάνα προηγουμένω, θέλουμε να δώσουμε λοιπόν αυτή την προσέγγιση, την σφαιρική, σε αυτό το συνολικό πακέτο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό το σημείο στην ανακοίνωση αυτή. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε τρει στόχου. Του ανέφερα, έχουμε όμω άλλου δύο. Καταρχήν, το να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει σε αυτό το πακέτο μεταρρύθμιση τα στοιχεία τα οποία εγώ θα ονόμαζα μη νομικά. Είναι προφανέ ότι τα νομικά κείμενα περιέχουν κάποιου περιορισμού. και νομίζω ότι οι περιορισμοί που συζητήσαμε πριν από λίγο ε, αντιπροσωπεύουν και μιλάνε σε βάθο για, για αυτούς τους περιορισμούς, αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μα το γεγονό ότι αυτά τα κείμενα είναι μη νομικά. Παρ' όλα αυτά, αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο τη μεταρρύθμιση. και το καλύτερο νομίζω παράδειγμα είναι ακριβώ η βελτίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Γι' αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Οπότε, για να βελτιώσουμε τι επιστημονικέ γνωμοδοτήσει, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι κάτι το νομικό. Βεβαίω υπάρχουν κάποια στοιχεία νομικά, όπω η υποχρέωση για συλλογή στοιχείων για τη βάση δεδομένων, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι βελτίωση τη επιστημονική βάση δεδομένων. Θα μπορούσε, α πούμε, να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των στοιχείων τα οποία δεν έχουν νομική φύση και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι και αυτά τα στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πακέτου. Θα θέλαμε λοιπόν να θέσουμε την ανακοίνωση αυτή υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα για να ζητήσουμε με τα όργανα. Υπάρχει ένας άλλος στόχος, ο εξής. Στα πλαίσια αυτής της, αυτού του σημαντικού πακέτου θα θέλαμε να τονίσουμε το ποιοι είναι για την Κομισιόν οι βασικοί στόχοι. Όταν ε, διαβάζουμε τα διάφορα στοιχεία και όταν ε, υιοθετείται αυτό το, αυτή η πρόταση από την ε, Κομισιόν είναι εύκολο να χαθεί κανεί στους μενάνδρους και στους λαβερίνθους, στους νομικούς. Να καταλάβει κανείς ακριβώς δηλαδή τι επιζητά η Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν τους στόχους μας να τους λέμε ξεκάθαρα όσον αφορά την Κομισιόν τουλάχιστον. Και η Κομισιόν λοιπόν προσπάθησε να συνοψίσει την μεταρρύθμιση σε αυτούς τους έξι μεγάλους άξονες, σε αυτούς τους έξι μεγάλους στόχους όπου θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αλευτικούς πόρους οι οποίοι θα διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο ώστε να περιορίσουμε τις απορρίψεις θα πρέπει να έχουμε μια μεταποιητική βιομηχανία η οποία θα είναι ανταγωνιστική και θα πρέπει επίσης να δώσουμε στην αλληλεία πιο ελκυστικές θέσεις απασχόλησης και με καλύτερες αμοιβέ. Θα πρέπει να θεωρήσουμε επίσης ως στόχο το γεγονός ότι ο τομέας της αλληλείας θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο αντίκτυπο στις παράκτιες οικονομίες και θα πρέπει να προσπαθεί να τις αναπτύσσει τόσο στον τομέα της αλληλείας όσο και στις συνοδευτικές δραστηριότητες της οικονομικής της αλληλείας γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικός στόχος για την αλληλεία να διατηρήσουμε μια σημαντική και ανταγωνιστική γεωργία για την Ευρώπη. Πέμπτο στόχο για την Κομισιόν είναι το να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα σημαντικό ρόλο στου Ευρωπαίου καταναλωτέ στα πλαίσια αυτή τη πολιτική μέσω αύξηση των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μα ώστε να επιτρέψουμε στου καταναλωτέ μα την ε, διεξαγωγή μια επιλογή όσον αφορά την αγορά των ψαριών που αγοράζουν και επιλέγουν και επίσης ότι θα πρέπει να πούμε ότι οι εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την αλληλεία συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για την Ένωση και αυτά θα πρέπει να διέπονται, αυτές οι δράσεις θα πρέπει να διέπονται από τους ίδιους στόχους που θέλουμε να εφαρμόσουμε στην κοινοτική μας αλληλευτική πολιτική. Ε, νομίζω, Πρόεδρε, συνοψίζοντας, αυτό είναι το περιεχόμενο και η στόχη αυτής της αναγκαίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πένια, αν συμφωνείτε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον ε, βασικό κανονισμό που σχετίζεται με αυτό το θέμα και μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πένια. Νομίζω ότι για τον βασικό κανονισμό να πω για άλλη μια φορά ότι αυτός ο κανονισμός βάσεις θα πρέπει να ειδωθεί υπό το φως αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή ότι αυτός ο κανονισμός παρέχει μία νομική βάση για την μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι σημαντικό για το μέλλον της αλληλείας περιλαμβάνεται εδώ και για τον εξή απλό λόγο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν είναι νομοθετήσιμα βάσει της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που θα έλεγα ότι εμπλέκονται και βρίσκονται πίσω από αυτή την πρόταση. Υπάρχουν όμω και πολλά άλλα στοιχεία για τα οποία δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε άμεσα και τουλάχιστον δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα με την τωρινή βάση τη κοινή αληθική πολιτική. Νομίζω ότι, όπω είπα πριν από λίγο, υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία σε αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσει τα οποία δεν έχουν νομικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, εσεί δεν θα τα βρείτε εδώ. Η βελτίωση, α πούμε, των επιστημονικών νομοθετήσεων δεν βρίσκεται εδώ. Και αυτό οφείλεται στο λόγο ότι ακριβώς δεν είναι νομικής φύσης αυτό το θέμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είναι εδώ. Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους του πακέτου μας. Να πω επίσης και το εξή. Θα ήθελα να περιγράψω αυτό τον κανονισμό και την πρόταση κανονισμού μιλώντας βάσει μια σύγκριση επιστημονική που έχουμε για την τωρινή αληθική πολιτική, όπου εντοπίζει ποια στοιχεία παραμένουν, ποια στοιχεία αλλάζουν κάπως και ποια στοιχεία στην ουσία είναι νέα σε αυτή την ε, πρόταση για την κοινή ελευθερική πολιτική. Νομίζω ότι σχετικά με τα στοιχεία τα οποία παραμένουν, πολιτικά δηλαδή στοιχεία τα οποία δεν αλλάζουν, θα πρέπει να μιλήσουμε καταρχήν για το θέμα των κανόνων πρόσβασης στα ύδατα το καθεστώς 12, μιλίων που όλες τι διαβουλεύσεις συμφώνησαν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο καθεστώς το οποίο γι' αυτό για μα δεν ήταν επιμαχό σημείο. Επίσης έχουμε το θέμα του καθεστώτος πρόσβαση στα ύδατα σε κάποια υπεράκτιες περιοχές. Εδώ εφαρμόζουμε το status quo και αυτό πάλι δεν αλλάζει. Μετά συνεχίζουμε με την ε, σχετική σταθερότητα η οποία ε, συνέλεξε διάφορε απόψει υπέρ τη διατήρησή τη στα πλαίσια τη διαβούλευση τη Πράσινη Βίβλου. Ούτε αυτό αλλάζει δηλαδή, ούτε επίση αλλάζει και το ότι θα χρησιμοποιούμε ως βασικό εργαλείο, παρόλο που δεν θα είναι αποκλειστικό ε, διαχείρισης ε, της ποσοστώσης, παρόλο που υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία υπέρ της διατήρησής τους, θα ήθελα να πω λοιπόν ότι παρόλο που διατηρούνται οι ποσοστώσεις ως βασικό στοιχείο, δεν κλείνουμε την πόρτα σε άλλες εξελίξεις, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, αν θέλουμε να πάμε σε άλλο σύστημα όσον αφορά την ευτική ικανότητα. Επίσης, διατηρούμε διάφορα άλλα στοιχεία του τωρινού καθεστώτος, όπως η δυνατότητα στα κρατημέλη να ευθετήσουν διάφορους κανόνες στα πλαίσια 12 μιλίων, η αδειοδότηση σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος γεωλογικός κίνδυνος κλπ. κλπ. Όλα αυτά, Πρόεδρε, είναι στοιχεία τα οποία δεν αλλάζουν για τον εξή απλό λόγο. Οι διαδικασίες διαβούλευσης είχαν ω εξή. Η Κομισιόν ε, δεν έβλεπε ότι υπήρχε λόγο αλλαγή όπω στην περίπτωση των 12 μιλίων ή σε άλλε περιπτώσει η Κομισιόν έβλεπε ότι ήταν ανοιχτή σε άλλε εναλλακτικέ λύσει. Όμω νομίζω ότι το αποτέλεσμα τη δημόσια διαβούλευση ήταν αρκετά ξεκάθαρο και υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία των χωρών μελών και του κλάδου και άλλων εμπλεκομένων που ήταν υπέρ της διατήρησης αυτών των στοιχείων. Αυτά, Πρόεδρε, συναψίζοντας κάποια από τα στοιχεία τα οποία δεν θα αλλάξουν κατά βάση. Υπάρχουν μετά κάποια άλλα στοιχεία της πολιτικής τα οποία θα αλλάξουν κάπως. Δηλαδή θα διατηρηθούν με κάποιες τροποποιήσεις. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Επί παραδείγματι το θέμα της διαχείρισης της ε, δυνατότητας του στόλου παραμένει όσον αφορά αυτά τα τμήματα του στόλου τα οποία δεν υπόκεινται στο σύστημα ποσοστώσεων, ίσως το σύστημα παραχωρήσεων, δικαιωμάτων κτλ. Ο λόγος είναι απλός επίσης. Η τωρινή πολιτική έχει νόημα όταν δεν υπάρχει κανένα εργαλείο το οποίο έχει αποδεχτεί ικανό να αλλάξει την δυνατότητα. Έχουμε το θέμα των παραχωρήσεων και των δικαιωμάτων που μέχρι τώρα αποδείχτηκαν ε, στοιχεία αποτελεσματικά όπου εφαρμόζονται. Οπότε θεωρούμε ότι από τη στιγμή που αυτά αποδείχτηκαν αποτελεσματικά δεν υπάρχει λόγος να καθορίσουμε μέγιστα όρια, τα οποία σε αυτή την περίπτωση θα ήταν περιτά. Κάτι το οποίο νομίζω εξάλλου αναφέρουν όλες οι αιτήσει εκθέσεις που αφορούν την πολιτική των στόλων. Υπάρχει επίσης το θέμα των ε, επιστημονικών νομοθετήσεων και τη συλλογή των δεδομένων για τις βάσεις. Υπάρχει μια ενίσχυση της υποχρέωσης των χωρών μελών όσον αφορά την παροχή δεδομένων για τις βάσεις όπως επίσης και υποχρέωση περιφερειακής συνεργασίας. Η κυρία Πατράων έβασε καμία ερώτηση προηγουμένω για το κατά πόσο δηλαδή εμεί επιθυμούμε διάφορε προτάσει οι οποίε περιλαμβάνονται στο πακέτο θα πρέπει να προσαρμόζονται και θα πρέπει να μπορούσαν να τροποποιηθούν ή να προσαρμοστούν σε μια μελλοντική αλλαγή προοπτική τη περιφερειακή πολιτική. Εδώ απλά και μόνο το ξαναλέω έχουμε να κάνουμε την ενίσχυση τη υποχρέωση των χωρών μελών για την παροχή στοιχείων για τη βάση δεδομένων. Αυτό θα συμπληρωθεί και είναι σημαντικό αυτό με μία σημαντική οικονομική ενίσχυση που θα αποφασίσουν χώρε μέλη για αυτό το στόχο. Οπότε δεν απαιτούμε απλά και μόνο νομικά από τι χώρε μέλη Εντάξει, απαιτούμε νομικά, αλλά βεβαίω έχουμε και οικονομική ενίσχυση όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων για τη βάση και αυτό επίση είναι τίμα λοιπόν τη πρόταση όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Επίση υπάρχει μια γενική, γενικότερη ενίσχυση του θέματο των ελέγχων και την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων στοιχείων της πολιτικής μας. Οπότε τι κάνουμε εδώ αν θέλετε, κάνουμε ένα είδος ε, αντίστροφης μηχανικής. Δηλαδή, κοιτάζουμε τις εξελίξεις που είχαν ε, οι έλεγχοι τα τελευταία χρόνια και οι κανονισμοί τους, σε σχέση δηλαδή με την νόμιμη αλληλεία, και τι κάνουμε. Λέμε ότι η νέα βάση της πολιτικής θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές τις νομικές εξελίξεις. Επίσης καθορίζουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με παραδείγματι με τα συμβουλευτικά συμβούλια, κατά το οποίο ήταν σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης του 2002, που θεωρούμε ότι παρόλο τους περιορισμούς τους ήταν ένα σημείο που σημείωσε επιτυχία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν και να εργαστούμε ώστε να τα βελτιώσουμε, τα συμβούλια, και θα θέλαμε λοιπόν να θεσπίσουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά την διάρθρωση αυτών των πεφριακών συμβουλευτικών συμβουλίων. Στη συνέχεια, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό που αποτελεί τα νέα στοιχεία, τα πιο καινοτόμα δηλαδή στοιχεία, τα πιο επίμαχα και τα πιο δύσκολα όμως επίσης της πρότασης αυτής. Καταρχήν έχουμε ένα στοιχείο το οποίο μας φαίνεται σημαντικό και είναι το εξής. Το να αφιερώσουμε μάλλον το να σωματώσουμε το νόημα της μέγιστης βιώσιμης ε, δυνατότητας στην νομοθεσία μας. Όπως ξέρετε υπάρχει αυτή η έννοια από το 2004-2005. Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε την ιδέα αυτή, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε βρει ιδιαίτερη θέση, κατάλληλη θέση στα νομικά συνοδευτικά κείμενα τη Αλία. Θέλω όμω να γίνει αυτό τώρα, γιατί πρόκειται για μια διεθνή υποχρέωση και ένα ξεκάθαρο στόχο της πολιτικής διαχείρισης, οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενσωματεθεί στη νομική βάση της αλίας, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Επίσης, επειδή, ε, μάλλον και αυτό δεν είναι νέο, αλλά αποτελεί ένα βήμα πρόοδου, είναι το εξή. Έχουμε τα πολιετή προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνονται στη νομική βάση την τοπική, αλλά με ένα νέο προσανατολισμό. Νέος προσανατολισμός, ώστε να πάμε βαθμια προς τα ε, συστήματα και τα συστήματα αλληλείας. Δηλαδή προσπαθούμε να απομακρυνθούμε έστω και τα θετικά από τα πολιτή διαχειριστικά προγράμματα που είχαμε μέχρι τώρα και όπως ξέρετε αυτά μέχρι τώρα ήταν ε, βασισμένα κυρίως σε ε, συγκεκριμένες, συγκεκριμένες μορφές αλληλείας. Αλλάζουμε λοιπόν τη βάση ώστε αυτά τα πολιτή προγράμματα να αποτελούν προγράμματα διαχείρισης τα οποία θα περιλαμβάνουν και θα σωματώνουν όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν. Θέλουμε δηλαδή να μετατρέψουμε τα πολυετή προγράμματα κατά κάποιο τρόπο σε βασικά εργαλεία περιφερειοποίηση τη κοινή αλληλευτική πολιτική και τη εφαρμογή, τη προσέγγιση για το οικοσύστημα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι κατ' ουσίαν νέα στην πρότασή μα. Επίση, νέο στην πρότασή μα είναι το να καθορίσουμε ένα ξεκάθαρο στόχο όσον αφορά την μείωση των απορρίψεων. Νομίζω, Πρόεδρε, να σας, ότι πρέπει να σα το εξηγήσω αυτό γιατί είναι από τα πιο δύσκολα και επίμαχα ζητήματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί η Κομισιόν ε, θεσπίζει αυτό το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υποχρέωση εκφόρτωση όλων αυτών των ειδών που έχουν εμπορικό ε, συμφέρον στην Ευρώπη. Ο στόχος του περιορισμού των απορρίψεων δεν είναι νέο. νέος. Το συζητάμε αυτό το θέμα εδώ και 5-6 χρόνια με άλλο επίτροπο που ξεκινήσαμε να βλέπουμε αυτά τα πράγματα και η εμπειρία στην Κομισιόν έδειξε ότι η προσέγγιση μας που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, δηλαδή το να κοιτάμε το θέμα αυτό από κάτω προς τα πάνω σε συνεργασία με τον κλάδο και τις χώρες μέλη και να δούμε ακριβώς τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν δυστυχώς, δυστυχώς εκτός από κάθε, κάποιες λίγες Θετικέ περιορισμένες εμπειρίες δεν έδωσε αποτελέσματα. Έδωσε αποτελέσματα τα οποία ήταν δυσκίνητα και ανεπαρκή. Οπότε τι έκανε η Κομισιόν. Προσπάθησε λοιπόν να μάθει από την εμπειρία άλλων χωρών, Νορβηγία και άλλων, όπου πράγματι προβλέπεται μια, ένας βαθμιός χαρακτήρας, μια διαβάθμιση, αλλά ακολουθήσαμε την εξή βασική προσέγγιση είχαμε μια υποχρέωση νομική για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και με βάση αυτή τη νομική υποχρέωση ξεκινήσαμε όλη τη διαδικασία διαβουλεύσεων ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το στόχο εφικτό. Θέσαμε λοιπόν την πολιτική πριν από την τεχνική ώστε να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα των απορρίψεων. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι το θέμα των απορρίψεων θα πρέπει να θυμίζεται μόνο από τι Βρυξέλλε όλε τεχνικέ λεπτομέρειε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, Πρόεδρε, και γι' αυτό ακριβώ η Κομισιόν θα ήθελε να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα είναι νομικά ε, δεσμευτικό για, την, για τον περιορισμό των απορρίψεων. Και από εκεί πέρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με την περιγραφή και τον καθορισμό τεχνικών, οικονομικών και άλλων στοιχείων, το οποίο θα μπορούσαν να μα βοηθήσουν στο να κάνουμε εφικτή την εφαρμογή αυτού του σημείου, τότε ευχαρίστως να ακούσουμε. Δεν έχουμε προκαταλήψεις δεν έχουμε βεβαίω ε, όλες τις λύσει στα χέρια μα. Είμαστε στη διάθεσή σα με κάθε διάθεση ώστε να ακούσουμε οποιαδήποτε καλή ιδέα για το πώ θα μπορούσαμε να κάνουμε εφικτό αυτό το στόχο. Πέραν τούτου, Άλλο ένα θέμα σημαντικό, η περιφερειοποίηση, θέμα το οποίο είχα την ευκαιρία και τη χαρά να συζητήσω εδώ στην ομάδα στο Κοινοβούλιο και το οποίο χαρίζει μια ε, ιδιαίτερη και συγκεκριμένη ε, παρατήρηση. Δεν χρειάζεται να επιμείνω για το όσον αφορά αυτό, αυτό το γενικό πτυχή της περιφερειοποίησης. Φυσικά και κάτι ισχύει σήμερα και έχει, κάποιο λόγο, διότι αυτό το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ενδιαφέρεται όσο γίνεται περισσότερο, τόσο ώστε να μπορέσει να φτιάσει μια τέτοια περιφερειοποίηση τη πολιτική. Και εμεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και βέβαια αντιλαμβανόμεθα 100% ότι το, το κείμενο είναι απογοητευτικό και επίση δεν μα δίνει ενδείξει για το τι μορφή θα πάρει στην αριστερά των μέλλον. Όμω υπάρχει κάτι άλλο, ότι αυτοί οι όλοι περιορισμοί είναι νομικής μορφής. Eh, Οπότε ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την καινούργια νομική βάση ε, λόγω της ε, συνήθειας της Όμως, πέραν αυτών των περιορισμών, υπάρχει ξεκάθαρα η δική μας η βούληση να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά για την περιφερειοποίηση. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία για αυτή τη συνεργασία και επίσης πιο συγκεκριμένα έχουμε όλα τα θέματα για τις λεπτομέρειες που θα οδηγήσουν ή στο να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ακόμα δεν, δεν έχει πάρει νομική μορφή, Όμω θέλουμε να το κάνουμε, θέλουμε να γίνει. Και οπότε και εμεί θα καταβάλουμε πάσα δυνατή προσπάθεια, θα συνεργαστούμε όσο γίνεται περισσότερο τόσο να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και αποτελεσματικά. Οπότε ε, σα επαναλαμβάνω ότι είμαστε ταγμένοι ω Κομισιόν ξεκάθαρα για να προχωρήσουμε προ την περιβιοποίηση. Και σα ε, επαναλαμβάνω, δεν είναι το ότι κάποια ε, ε, πράγματα δεν έχουν λάβει νομική μορφή, δεν τα λέει ο νόμος του και ότι δεν συμβαίνουν. Γιατί πολλά, πολλά μπορούν να γίνουν. Οφείλουμε να τα κάνουμε και ακριβώς ε, είναι δυνατό να, τους, ε, να τα πρικοδοτήσουμε αυτή την νομική βάση. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με τις επιστημονικές νομοδοτήσεις, γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και αυτό και όλοι προς τα εκεί κοιτάμε. Τώρα κάτι άλλο τελείως καινούριο είναι το ότι θέλουμε να συγκροτήσουμε ένα σύστημα με κάποιο είδου ε, άδειε ε, μεταβιβάσιμες σε σχέση με τα μικρά ελευτικά σκάφη. Και αυτό το προτείνουμε διότι, κύριε Πρόεδρε, όταν εσείς ε, ρίξετε μια ματιά σε αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, βεβαίω εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω το τι θα αποφασίσει, τι θα κρίνει το ελεγκτικό συνέδριο, όμως Ακριβώ μια που υπάρχει διαφάνεια στι εργασίε μα, έχουμε μια ιδέα ότι γίνεται μια που υπάρχει διαδικασία διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μυστικό αυτό ότι το Ελληνικό Συνέδριο πριν γνωμοδοτήσει έρχεται σε επαφή μαζί μα. Και ακριβώ και γι' αυτό κάποια ιδέα έχουμε, έστω και γενική. Οπότε, ε, όπω λέμε, ξέρουμε κατά πού θα πάνε, τι κατεύθυνση θα πάρουν τα πράγματα. πού το πάνε λοιπόν θέλουν να πούν ότι η σημερινή πολιτική για τον ελευτικό στόλο έχει δύο σημεία επί των οποίων επικρίνεται σφόδρα. Δηλαδή βασίζεται σε κάποιες σταθερές παραμέτρους που δεν αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο. Οπότε μιλούμε για μια πολιτική που ελέγχεται από αυτές τις παραμέτρους ε, γιατί ας πούμε είναι ο κινητήρας και υποδύναμη όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες του σημερινού αλευτικού στόλου. Άλλο στοιχείο, ε, προφανές, αυτό το οποίο και εσείς μας αναφέρατε, ότι δηλαδή η πολιτική στήριξη για την επίλυση του προβλήματος βασίζεται σε αυτές τις απορρίψεις. Ε, αυτό γίνεται παντού. Όλοι έχουν κάνει μειώσεις, αποσύρσεις και τελικά διαπιστώνουμε ότι έχουμε δαπανίσει τόσο προχρήματα φορολογουμένων χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Πρόβλημα που δεν μπορεί να γνωρίσει η Επιτροπή. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Ήδη αυτά τα αποπειραθήκαμε στο παρελθόν, συγκεκριμένοι στόχοι ανακρατός μέλλον και τελικά δεν ε, υποχρεώνουμε κανέναν να καταργεί, να παροπλίζει πλοία. Και μετά να πηγαίνουμε και να δίνουμε και χρήματα. Όμως είπαμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο μέσο αποτελεσματικό για να γίνει μεταρρύθμιση στην Ελία. Οπότε αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο που ε, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γίνεται αποπολιτικοποιημένα. Μην έχει φόρτιση η πολιτική. Η πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό. μόνο γιατί μας λένε ότι έχουμε αιμονή στο να παραπλήσουμε πλοία. Όχι, με τίποτα δεν ισχύει αυτό. Ο κλάδος να το αποφασίσει. Ακριβώς αυτό το μέτρο. Αυτοί να αποφασίσουν τι θεωρούν οι ιδιώτες όσον αφορά αριθμό σκαφών για να κάνουν τη δουλειά τους. Φάνηκε. Ότι με αυτή τη μέθοδο κάτι κάνουν για να επιλύσουν το πρόβλημα. Και επίσης τα κράτη-μέλη και μέρος του κλάδου έχουν κάποιες επιφυλάξεις, κάποιους φόβους όσον αφορά ε, αυτό το μέσο πολιτικής. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι τα κράτη-μέλη δίνανται να θεσπίζουν μια ολόκληρη σειρά μέσων, τόσο ώστε να περιορίζουν τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα. Να έχουν δηλαδή λίγοι, για παράδειγμα, πάρα πολλά ελευθερικά δικαιώματα. Μπορούν τα κρατημέλη να βάζουν όρια σε σχέση με αυτές τις άδειες. Άρα, έτσι μπορεί και τα κρατημέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο και αν έχουν και αυτές τις, ας τις πούμε, ρήτρες διαφύλαξης, ούτως ώστε αυτά τα πιθανά ε, αρνητικά σημεία, αυτούς τους θεμητούς φόβους να τα αντιμετωπίζουν. Επίσης, Πρόεδρε, υπάρχει ένα κεφάλαιο όπου για πρώτη φορά για αυτό και το βάλουμε λέει ότι θα πρέπει η πολιτική μας γενικότερα να έχει κοινούς στόχους. Είπαμε δυναμική πολιτική θα πρέπει οι πολιτικές μας ε, η μία με την άλλη να έχουν συνέπεια. Επίσης για την ηχθειοκαλλιέργεια έχει ένα κεφάλαιο που μέχρι τώρα δεν προβλεπόταν στα κοινωνικά κείμενα. Έχουμε συμπεριορισμένες αρμοδιότητες για την ε, ηχθειοκαλλιέργεια, όμως θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά με κάποιο οικονομικό μέσο την εχθροκαλλιέργεια. Όμως δεν θα πετύχουμε τίποτα, θα πετύχουμε πάρα πολύ λίγα εάν τα κράτη-μέλη υπό την εθνική αρμοδιότητα δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν τόσο ώστε να δώσουν μια όθηση στη Γεωργία. Άρα χρειάζεται διοικητική απλούστευση να διευκολυνθεί επίσης η πρόσβαση στο χώρο, να αρθούν κάποιες αντιφάσεις όσον αφορά την χρήση θάλασσας και ξηράς υπό την, ε, στην μάλλον εθνική επικράτεια. Έρευνα και οικονομική ενίσχυση δεν αρκούν, διαπιστώθηκε. Άρα, θα πρέπει να έχει μάθει το μάθημά του το κάθε κράτο μέλο ώστε να μπορεί να δώσει μια όθηση στον τομέα τη χειροκαλλιέργειας. Επίσης θα βάζουμε και μια νομική βάση που δεν προβλέπεται μέχρι σήμερα και λέει με ποιες αρχές πρόκειται να οργανώνεται η, η κοινή οργάνωση της αγοράς. Και όπως ε, ξέρετε έχουμε κάποιες, ε, κάποιους στόχους, κάποιες αρχές που επίσης τώρα έχουν ε, αναπτυχθεί επί τη βάση του χρηματοοικονομικού μέσου που, θα προβλέπεται. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό για τη γνώμη μας είναι το να υπάρχει μια ξεκάθαρη νομική βάση. Και έτσι να καθορίζεται το πώς θα γίνει, υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις η χρήση των πόρων. Μέχρι σήμερα με τα επιχειρησιακά προγράμματα παίρνουν τα κρατημέλη το κοινωτικό χρήμα. Όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει το ότι αυτοί οι οικονομικοί πόροι δεν δαπανώνται απλώς μόνο με μια χρηστή διαχείριση αλλά και ότι δαπανώνται με τρόπο που να βοηθούν στην επιτυχία των στόχων γιατί σήμερα δεν έχουμε ένα τέτοιο τρόπο. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ότι το χρήμα του φορολογουμένου Ε, πηγαίνει σε κινήσεις που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων. Βεβαίω αυτό θα, θα πάρει και νομική μορφή, ότι δηλαδή αυτοί οι πόροι θα πρέπει να βοηθούν στην επίτευξη των στόχων. Και έτσι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσο θα εκταμιεύσει αυτού του ε, πόρου. Άλλωστε, ε, αυτά όλα δεν είναι καινούργιο τελείω γιατί είναι στοιχεία τη κοινή αγροτική πολιτική και αλλού. Και τώρα θα είναι και ένα στοιχείο καινούργιο τη ελληνική πολιτική. Να λοιπόν τι δεν άλλαξε καθόλου, τι άλλαξε ελαφρά και τι στοιχεία είναι όλο. Ναι. Εμεί ευχαριστούμε λέει πρόεδρο. Και τώρα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα για αυτό το χρονοδιάγραμμα. Όπως τα εξήγησε ο εισηγητής. 11 μήνες. Αυτό είναι ε, με κριτήρια οποιοδήποτε κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ αργά. Για πρώτη φορά ξέρουμε ότι τα κοινοβούλια θα βοηθήσουν στην αναθεώρηση. Και πολλές φορές λέμε, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία. Τελευταία ευκαιρία να σώσουμε τις θάλασσες. Άρα, επομένω, ελπίζω ότι αυτό το χρόνο το χρησιμοποιήσετε ε, δημιουργικά και θα καταλήξετε σε κάποια διακομματική συμφωνία και να προχωρήσουμε μια τέτοια μεταρρύθμιση, ούτω ώστε να μπορούμε να επηρεάσουμε το τελικό πακέτο. Για την Κομισιόν έχουμε εδώ πέρα μια σειρά στοιχείων του βασικού κανονισμού που δεν προκύπτει ότι θα αποδώσουν όσον αφορά τη διαχείριση και το σχετικό πρόγραμμα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει έτσι όπως σιγά σιγά εκπονεί τον, ε, το νέο κείμενο, θα μπορέσει να άρει κάποια κενά που υπάρχουν μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόση επιστημονική πρόοδο, ακόμα έχω μεγάλα κενά. Δεν καταλαβαίνω γιατί η επιστημονική μας τεκμήριωση ε, είναι τόσο ελληματική μετά από τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει. Και πώς και με πόσα χρήματα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δουλεύουμε επί τη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Θέλουμε το 2015 να έχουμε όσο γίνεται το, το, το, το, το, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αλλά είπαμε ότι με το 2030 δεν θα χειροκροτηθεί η μεταρρύθμιση. από την άλλη μεριά βέβαια, να μην έχουμε υπεραλίευση. Δεν φαίνονται τόσο φιλόδοξες προτάσεις Κομισιόν. Στοχεύουν στο να υπάρχει επαρκή πόρων και έτσι να υπάρχει υψηλή απασχόληση και επίσης επάρκεια τροφίμων. Για, τη... για την ελία μικρής κλίμακας είπαμε ότι είναι το 10% της απόδοσης του ελιεύματος και είπαμε ότι θέλουμε να είναι με βιώσιμο τρόπο να υπάρχουν ψάρια. Και αναφέρεται ότι τα σκάφη αναλόγω το μέγεθό του θα υπάγονται όχι στο καινούριο πρόγραμμα. Αφού όμως αυτού του είδου η αλληλεία μα δίνει πόρου και απασχόληση, τι θα βρεθεί για το μέλλον σαν κίνητρο. Πολλές γνώμες έχουν ακουστεί. όλα τα θεμητά παράπονα ή αιτήματα θα πρέπει να καλυφθούν. Και επίσης την υπεραλίευση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπω είπατε και εσεί πρόεδρε. Άρα, απόκειται σε εμά αλλά και στα κρατημέλη και στου αλλιεί, να δούμε το ότι πάρα πολύ εύκολα επικρίνει κανεί τις προτάσεις αλλά θα πρέπει να δεν αρκεί να πει τι δεν του αρέσει θα πρέπει να πει τι θέλει. Επομένως πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ελευθερικές δυνατότητές μας, με τα TFC θα βρούμε μια λύση. Αν όχι, να βρεθεί μια εναλλακτική. Ευχαριστώ, ε, ε, Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, όσον το χρονοδιάγραμμα. Και εγώ έχω φτιάξει ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα για την κοινή οργάνωση αγορά ή το CMO τέλος πάντων και θα πρέπει να δει η Επιτροπή σαν μια συνέχεια της ε, μεταρρυθμίσης όπως και θα πούμε και αργότερα οπότε καλύτερα ε, να περιμένουμε και αργότερα να δω καταφέρουμε γίνεται περισσότερα γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι εκθέσεις εάν πάνε σε τρία ανάγνωση και σε τριγωνικό διάλογο θα πάνε για 18 μήνα. Άρα θα έχουμε φτάσει μέσα του 2013 για να έχουμε προχωρήσει. Και εγώ σήμερα υπέβαλα τρία ερωτήματα στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας απασχολούν πριν αρχίσουμε να κατεβάζουμε κάποιες τροπολογίες για το πακέτο συνταρρυθμίσεις. Οπότε έχουμε εδώ τρία βασικά θέματα. Περιφερειοποίηση, μεταβιβάσιμες άδειες αλίας και το τρίτο είναι οι απορρίψει. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκχωρεί στα κρατημέρη τη δυνατότητα να δρουν αντί για εκείνη Για διάφορα θέματα. Άρα χρειάζεται όμω να ξεκαθαριστεί στην πράξη αυτό πώ θα λειτουργεί. Πώ θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια περιφερειοποίηση που να έχει νόημα. Κάτι το οποίο πάντοτε το θέλαμε όσον αφορά το πακέτο της μεταρρύθμισης. Αυτό το οποίο θέλει η Επιτροπή είναι να έχει ένα κουτί με εργαλεία και να, να διαλύει το κάθε κράτος μέλος ό,τι είναι πιο κατάλληλο για να κάνει τη διαχείριση των ελευτικών πόρων. Να κάνει ό,τι γίνεται τώρα για τα TFC. Επιτρέπεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμένει σε τέτοια μέτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Και αυτό σε κάποια κρατημέλη να αποβαίνει παραβίαση συνθήκης. Θα ήταν θεμητό και νόμιμο να ζητηθεί εθελοντικά να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Γιατί και αυτές οι άδειες αλίας είναι πολύτιμο μεσοπολιτικής. έχω μιλάμε για μια δεκαπενταετία. Βεβαίω και οι μεγάλες εταιρείε θα ζητήσουν τέτοιε συγκρίσει. Δεν θέλουμε όμω να υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση στα χέρια λίγων γιατί αυτό θα αποσταθεροποιήσει την αλληλεία σου. Και όσον αφορά τις απορρίψεις, τι θέλει ο Ευρωπαϊκή θέλει να αλλάξει το ισχύον δίκαιο. Όταν κάποιο λοιπόν εκφορτώνει κάποια ψάρια μικρά, μικρού μεγέθους, εκτός ποσόστοσης, αυτά τι θεωρούνται. Από ό,τι έχω κατάλαβα από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή και θα παραμείνει παραμαλίευμα. Να το δίλημα που έχει ο ψαράς. Αναγκάζεται να εκφορτώσει παραμαλίευμα. Είναι βέβαια και οικονομικό το θέμα. Αυτά κανονικά θα είχαν απορριφθεί είναι βασικά ερωτήματα που ελπίζουμε η, το, το, η νομική υπηρεσία θα δώσει απαντήσεις. Και έτσι θα ξέρουμε τι ισχύει πριν υποβάλουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σχόλια τώρα σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Καταρχήν, ε, το, αυτό που έχει να κάνει με την πρόσβαση, με τον, με τον κανόνα αυτό και για τη ζώνη των 12 μιλίων. Η Επιτροπή λέει ότι κάνει ένα απολογισμό μάλλον θετικό. Έχουμε ένα θέμα στο οποίο φαίνεται ότι πολλοί να συμφωνούν. Σίγουρα υπήρξαν θετικές εμπειρίες με τον ορισμό ε, για την ε, ε, πρόσβαση στα 12 μίλια. Επιτρέπει το θέμα του συνδυασμού της αλίευσης σε σχέση με τις παράκτιες ζώνες. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει σίγουρα το συντονισμό και όλα αυτά που λέγονται και συμφωνώ. Αλλά το ερώτημα μου είναι το εξή. Και γιατί όμως διατηρείται σαν εξαίρεση και δεν μεταφράστηκε σε κάτι οριστικό. Εξάλλου, κάτι άλλο. Γιατί να μην αυξηθεί αυτή η αποκλειστική ζώνη για πρόσβαση. Διότι θα μειώνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο πίεση όσον αφορά τους σπόρους διότι είχαμε μέχρι τώρα πίεση πάνω στο θέμα των αποθεμάτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι θετικό. Να δοθεί μια πιο οριστική ρύθμιση πάνω σε αυτό το θέμα. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας ε, όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γυτνίαση. Η Επιτροπή μας λέει ε, ότι η συμφωνία εν μέρει λοιπά, Αλλά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τη συνθήκη. Τώρα, για τις ελλείψεις όσον αφορά τις ε, γνώσεις όσον αφορά την επιστημονική πτυχή. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κεντρικό θέμα του διαλόγου μας. Όταν υπάρχουν ε, ε και χαίρομαι που το αναγνωρίσει η Επιτροπή, αλλά πριν από, λίγες, ε, πριν από λίγους μήνες έχασε μια ευκαιρία η Επιτροπή όταν συζητήσαμε τον κανονισμό εδώ στο Κοινοβούλιο και εγώ ήμουν εισηγητής. Και, και εγώ τι έλεγα, αύξηση τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δράση, στη χρηματοδότηση των δράσεων όσον αφορά για να, την επίτευξη δεδομένων πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί έχασε λοιπόν πριν από μήνες αυτή την ευκαιρία η Επιτροπή. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επιβαρυθούν επιπλέον τα κράτη-μέλη λέγοντάς τους ότι εσείς θα πρέπει να πετύχετε να συλλέξετε περισσότερα δεδομένα. Στις χώρες μας τώρα, τι κάνουμε, έχουμε προβλήματα, κλείνουμε νοσοκομεία, σχολεία, ε, τα δημόσια, οι δημόσιοι πόροι μειώνονται και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τι λέτε, τι μας λέτε, να έρθουν οι χώρες μέλη να αναλάβουν επιπλέον χρηματοδότηση για να συλλέξουν δεδομένα για τις αποκλειστικές ζώνες. Θέλετε δηλαδή να επιβαρηθούν επιπλέον οι χώρες μέλη. Πρέπει να εξασφαλίσετε ε, χρηματοδοτήσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Ρωτά λοιπόν ξανά. Γιατί άφησε να περάσει αυτή η ευκαιρία η Επιτροπή πριν από λίγους μήνες. Τώρα, για την κατάργηση όσον αφορά την απόρριψη αλευμάτων. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ψυχές οι οποίες δεν είναι νομικής φύσεως και είναι σημαντικές για αυτό το πρόβλημα. Ζητάω από την Επιτροπή να μας πει, έχει σκεφτεί κάποιες λύσεις πέρα από τον ορισμό ενό χρόνου διαγραμμάτων. Έχει σκεφτεί κάποια λύση για να πετύχει τους στόχους αυτούς, ξέροντας ότι ένα μεγάλο μέρος των απορρίψεων έχουν να κάνουν με την, με την εμπορική διάσταση. Τι σκέφτηκε πάνω σε αυτό το θέμα η Επιτροπή, δηλαδή με τη, σχέση με την εμπορική διάσταση. Τώρα, για, τον, ε, για τα δικαιώματα τα μεταφέρσιμα. Και εδώ πάλι τα ίδια έχουμε. Μια παρατήρηση. όταν έχουμε με κάποια περιοριστικά συστήματα. Αυτά μας φέρνουν σε, δημιουργούν μια αντίφαση σε σχέση με τη θέληση που έχει εκφράσει η Επιτροπή να υπάρχει μια αποκεντροποίηση. Τώρα έχουμε μια τάση αντίστροφη. Έχουμε εμπειρίες και από άλλες χώρες, τρίτες χώρες μάλιστα, όπου διαπιστώνει κανείς ότι ε, υπάρχει ένας τρόπος ε, αυτό είναι ένας τρόπος πολύ αποτελεσματικός για να μειωθεί ο αλλιευτικός στόλος. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε διότι έχουμε ένα διάλογο που επικρατεί στην, Ευρω... στην Επιτροπή όπου ε, το... η κατευθυντήριος γραμμή είναι να ανοίξουμε τα πάντα στην αγορά. Η αγορά θα ελέγχει τα πάντα. Βλέπουμε όμως ποιες είναι οι επιπτώσεις στις χώρες που γίνεται κάτι τέτοιο. Γίνεται ένα συγκεντρωτισμός, μείωση ε, ε, αλληλευτικού στόλου, ε, πλήττονται, πλήττονται οι, παρα, οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή αλληλεία. Ρωτώ λοιπόν στην Επιτροπή, ότι έχει υπάρχει μια ε, ρήτρα εδώ και πώς μπορείτε να φανταστείτε ότι με μια ρήτρα έτσι ως για μαγεία θα μπορέσετε να αποκλείσετε ένα συγκεντρωτισμό σε αυτόν τον τομέα. Η Επιτροπή λέει ναι, ναι, συμφωνεί ότι όσον αφορά την περιφερειοποίηση και μετά μας λέει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ρωτώ λοιπόν στην Επιτροπή, αυτή η ρήτρα που αναφέρατε, πώς θα έρθει, ας πούμε, πώς θα είναι συμβατή με την συνθήκη της Λισαβόνας. Πώς θα γίνει δηλαδή, από τη μια έχουμε τις αρχές της συνθήκης, μιλάμε για ελεύθερο ανταγωνισμό, Δεν θα μας πείτε δηλαδή ότι μην ανησυχείτε για τον συγκεντρωτισμό που μπορεί να υπάρχει στον τομέα, θα εξασφαλίσουμε κάποιες ρήτρες, κάποιες εξαιρέσεις. Είναι δυνατόν. Όντως η συνθήκη, η συνθήκη λέει ότι όλες οι ρήτρες για εξαιρέσεις θα πρέπει να υποτάσσονται στον ελεύθερο ανταγωνισμό, στην ελεύθερη αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα και αν μιλάει κανείς για εθνικά συστήματα, αναπόφευκτα θα υπάρχει ένα συγκεντρωτισμό σε ε, κοινοτική κλίμακα. Διότι αυτό που λέει, αυτό το λέει η συνθήκη της Λισαβόνα. Όλες οι ρήτρε, εξαιρέσεις κλπ. θα ε, υπόκεινται ε, στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ. Ησυχία. Κύριε Μιλάνα. Σύντομος θα είμαι. Νομίζω ότι θα πρέπει να γραφτεί από την αρχή η μεταρρύθμιση. Να μου πει Κομισιόν, αν το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να υιοθετήσει αυτή τη διάταξη, όπως ακριβώς μας την παρουσιάζεται, και αυτή η διάταξη μετατραπεί σε νόμο, τι ακριβώς θα βελτίωνε, τι αλλάζει όσον αφορά την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που ήδη συμβαίνουν, δηλαδή η θάλασσα ήδη συνεχίζει να μην έχει την δυνατότητα αναγέννησης και οι άλλοι έχουν όλο και λιγότερα αλλιεύματα προς αλλιεύση. Νομίζω δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο στου επόμενου 11 μήνε να γίνει η μεταρρύθμιση. Και από το Κοινοβούλιο. Όμω έχω την εντύπωση ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι είδο προσαρμογή τη πορεία, εμπλό δηλαδή, κανόνων που αποδείχτηκαν περιορισμένοι και κατέδειξαν τα όρια τους όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν ε, περιμένω θαύματα. Να πω μόνο ότι συμμερίζομαι την ιδέα ότι τα δικαιώματα δεν γίνεται να παραχωρούνται. Συμμερίζομαι την ιδέα και την αρχή ότι ίσως να χρειαστεί να αλλιεύουμε λιγότερο και να αλλιεύουμε όλοι μας. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ μικρής και μεγάλης κλίμακος αλίας. Συμμερίζομαι επίσης την ιδέα ότι η αλλιά πρέπει να είναι ένα κοινό αγαθό δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι μεγάλες προκλήσεις να περιλαμβάνονται. Δεν βλέπω να περιλαμβάνονται σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Έχουμε ένα μοντέλο το οποίο προβλέπει και προτείνει προσαρμογές στο τάδε ή δινά σημείο και μετά μετά από κάποια χρόνια θα λάβουμε υπόψη μας τις κριτικές οι οποίες θα ασκηθούν σε σχέση με τις υπέρμετρες δαπάνες που θα γίνουν και οι οποίες δεν θα έχουν θετικά αποτελέσματα ε, και θα ξαναγυρίσουμε έτσι και θα ξανα προσαρμόσουμε την πολιτική μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες. Νομίζω ότι η συζήτηση στο Κοινοβούλιο εκτός από δυσκίνητη και έντονη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει την πρόταση αυτή. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση αυτή της ε, Κομισιόν είναι ανεπαρκής όσον αφορά την προσέγγιση της, δηλαδή η προσέγγιση της Κομισιόν η οποία κάνει μικροπροσαρμογές, ρεμέτια δηλαδή. Να πω και κάτι τελικό. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Λείπει όμως μια συνολική πολιτική. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση χωρίς πνοή. Γιατί δεν προσφέρει στη συζήτηση για το κλάδο μια έστω ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Ίσως εδώ να υποτιμάμε το εξή. Υπάρχει μια θάλασσα στην οποία υπάρχουν όλο και λιγότερα ψάρια και υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος έχει τεράστιες επιπτώσεις οικονομικές λόγω της έλλειψης αλλιευμάτων. Νομίζω ότι ο μηχανισμός που μας υποβάλλεται για έγκριση δεν υπάρχει καμία ένδειξη λύσης προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ για το στόχο μέσα με τον κύριο Ντέβις. Είπαμε ότι συμφωνούμε. Φαίνεται βέβαια δύσκολο να επιτευχθεί ε, με χρονικό το 2015. Όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το MSY δεν είναι μόνο τρόπος υπολογισμού των ελευθερών πόρων αλλά και της εθνισμότητας. Άρα, αύριο θα μπορούσαμε να ξέρουμε. Από ξεκαθορίσουμε τι στόχο βάζουμε όσον αφορά τη θεσιμότητα. Άρα, ας μην απογοητευόμαστε. Επίσης, για κοιτάξτε για τη Βαλτική, τι έχει πει ο οργανισμός σα. Τι γίνεται εκεί με το βακαλάο. Ε, αν ακολουθήσουμε το, το, MSY, τότε πάμε για μεγαλύτερε ποσοστέ του χρόνου. Σε σχέση με τη μακρόπνα διαχείριση. Μιλάμε για αύξηση 15% ετησίως, οπότε έτσι εκεί το απόθεμα θα αυξηθεί πολύ περισσότερο από όσο να είχαμε καθαρό καθεστώς MSY. Και επομένως έτσι θα είχαμε μακρόπνοη βιωσιμότητα, αυτήν την οποία επιδιώκουμε. Άρα Ίσως ε, το MSY δεν είναι αρκετά φιλόδοξο, επομένως ε, πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο σας είπα για, να είμαστε πιο σωστοί όσον αφορά και το περιβάλλον και το απόθεμα. Τώρα, όσον αφορά τις απορρίψεις, να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να έχετε στη λίστα σας ε, κάποια εμπορικά ψάρια και λέτε ότι πρέπει να υπόκειται τις απορρίψεις. Όχι δεν είναι ούτε πουλιά, ούτε θηλαστικά. Ε, τι θα κάνει, θα γίνουμε με, με τα υπόλοιπα ψάρια. Απαγόρευση, απόρρευση είναι απαγόρευση, απόρρευση. Όπως κάνουν οι Νορβηγοί, Ισλάνδοι. Δεν είναι δυνατόν. αν δεν τα αναφέρετε, αν δεν αναφέρετε τα είδη που θέλετε, πώς θα τηρηθεί η απόγρευση. Τώρα όσον αφορά το οικονομικό φρούτο της συμφωνώ με τον κύριο Στίβενσον. Ναι, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οι πόροι που περισσεύουν τις ποσοστώσεις, πώς θα χρησιμοποιηθούν, τι θα γίνει με την ποσόστοση για τις απορρίψεις, αν θέλουμε να έχουμε μια νέα αγορά για τα είδη που υπόκεινται την απόρριψη. Για να δούμε πώς θα μπουν στο σύστημα ελέγχου ε, τα, τα, τα ωφελήματα, ό,τι τέλο πάντων προκύπτει από την απόρριψη. Να πάνε, ξέρω εγώ, σε ακτοφυλακή κλπ. Για την περιφερειοποίηση τώρα. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα στην πρόταση. Ε, ήδη μα έχει δώσει επεξηματικό κείμενο. Μα έχει υποσχεθεί μάλλον υποσχεμένο κείμενο η Κομισιόν Κάποιε προτάσει για αυτά τα κοτιά εργαλείων. Και με αυτήν την εργαλεία τέλο πάντων τα κρατημένα θα εφαρμόσουν την περιφερειοποίηση, οπότε ε, η συζήτηση θα στηριχθεί εκεί πέρα. Τώρα όσον αφορά τα TFC. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Στίβενσον σε σχέση με την νομιμότητα της επιβολής των ε, TFC στα κρατημέλη. Αυτό είναι σύνομο σε σχέση με την συνήθεια της Λισαβόνας. Μιλάμε δηλαδή για χρησιμοποίηση των, ε, των φυσικών πόρων. Μπορεί να κάνει το στα κρατημέλη επίσης Τα κράτη-μέλη σε κρατικό, σε εθνικό, σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ενεργήσουν άπαξ όμως και τα δικαιώματα έτσι όπως έγινε στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί λανθασμένο όσον αφορά τις αδειοτήσεις να βρεθεί ένα σύστημα κατά το οποίο θα παραχωρούνται οι αδειοδοτήσεις προς εκείνους που από πλευρά ε, κοινωνική και περιβαλλοντικής ψαρεύουν με τον πιο φιλικό τρόπο, τον πιο βιώσιμο τρόπο. μας τα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν ανοίξει κανένα θάλασσα. Ελεύθερο είναι όποιο θέλει να πάει και να ψαρέψει. Αυτό είπαμε ότι είναι η θεμελιώδης αρχή της αλίας. Αλλά τώρα να ιδιωτικοποιήσουμε του ωκεανού και να πούμε όχι, πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία. Ποσόστοση. Γίνεται αυτό. Μα τα ψάρια ανήκουν σε όλου. Είναι κληρονομιά κοινή τη κοινωνίας και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η βασική αρχή και δεν είναι δυνατόν να παραχωρήσουμε αυτά τα δικαιώματα. Για ποιο χρονικό διάστημα. Να υπάρχει ένα σύστημα λύση, λύση τέλος πάντων, κατά το οποίο πληρώνει κανεί το κράτο για να πάρει την ε, έγκριση, την άδεια και το κράτος χορηγεί στους καταλληλότερου την άδεια να ψαρέψουν. Κύριε Γκάλγαρη, επειδή είχατε φύγει δεν σα. είδα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η γενική συζήτηση σήμερα το πρωί, έστω και αν ξύσει το κόπο, να πω ότι χαίρομαι, έστω και αν έχω επιφυλάξει που ακούω την Κομισιόν να τα αποστηρίζει όλα αυτά Είναι σημαντικό λοιπόν και εμείς να υποστηρίξουμε τον κύριο Στίβεσον και την νομική παροχή, την νομική γνωμοδότηση που μας παρήχε σε σχέση με την περιφερειοποίηση. Ίσως θα πρέπει να πούμε ότι εμείς είμαστε έτσι μη τεχνική σε σχέση με τα νομικά θέματα εμείς και θα πρέπει να πούμε ότι για την περιφερειοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει στην πράξη, όχι ιονή. Με τον κατάλληλο τρόπο βέβαια. Και χαίρομαι που ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε σήμερα θα πρέπει να γίνει περιφερειοποίηση, οπότε εντάξει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα πετύχουμε τελικό αποτέλεσμα, να βρούμε έναν τρόπο και να δούμε ποιος άλλος μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Να πω ότι χάρηκα πολύ που είδα για την επέκτηση των ορίων. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο όλες οι χώρες θα συμφωνήσουν γιατί οι χώρες οι οποίες ήταν πιο προκλητικές ε, έχουν μαζέψει τα πιο πολλά ψάρια από τις θάλασσες οπότε δεν ξέρω η ιδέα είναι καλή βεβαίως αλλά θα έπρεπε να την επεκτείνουμε αυτή την ιδέα ώστε να καταστεί αυτό κάτι το θετικό για τη βιωσιμότητα των αλευμάτων για τα επιστημονικά δεδομένα. Ναι, βεβαίω, είναι σημαντικά αυτά, όπω και οι επιστήμονε. Υπάρχει όμω άλλο ένα στοιχείο εδώ, οι εμπλεκόμενοι και οι διάφοροι Θα πρέπει να υπάρχει συνεχή ανταλλαγή απόψεων με του εκπροσώπου των εμπλεκόμενων, των εμπλεκομένων στον τομέα τη αλληλεία. Επειδή αυτοί έχουν μεγάλο λόγο, έχουν σημαντικά πράγματα να μα πούνε. Εκτός δηλαδή από τη συμμετοχή τους, η οποία είναι η τεχνική, η κανονική, η επαγγελματική σε ημερησία βάση, έχουν και απόψεις σε σχέση με την πολιτική, οπότε θα πρέπει να τους ακούμε πάντοτε. Ε, και σχέση με τα επιστημονικά δομένα και σχέση με όλο, όλες τις εξελίξεις στον τομέα. Και κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα υπέρ της παραχώρησης ή της μεταβίβασης μεμονωμένων ποσοστώσεων. Η αγορά των δικαιωμάτων δεν νομίζω να βοηθήσει και τόσο τα λίευματα και τα λευτικά αποθέματα. Ίσως το αντίθετο. Και σήμερα το πρωί να πω ότι είχαμε μια συνάντηση σε σχέση με ένα ενδεχόμενο ψήφισμα ώστε να κάνει το, το, το κείμενο πιο ισορροπημένο, αλλά να πω ότι αυτή η άποψη που άκουσα προηγουμένω ήταν η πιο ακραία, η πιο δεξιά σε σχέση με, με την αλία. Και νομίζω ότι η απλότητα του επιχειρήματο στην, στην ουσία μας, μας προκαλεί να αντιδράσουμε έχουμε επιχειρήσεις της Ισπανίας που έρχονται και αλλιεύουν στην Ιρλανδία. Εμείς λοιπόν δεν γίνεται να το επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Και μετά ας υποθέσουμε προς στιγμή ότι αυτές οι παραχωρήσιμες ποσοστώσεις εφαρμόζονται. Εδώ αυτό θα έχει διακρίσεις σε αυτούς που αλλιεύουν με διαφορετικό τρόπο, αλλιεύουν παράκτια κλπ. Τι θα κάνουν λοιπόν αυτοί. Δεν θα, μείνουν, θα μείνει τίποτα. Θα τα λείψουν όλα οι άλλοι και θα αναγκαστούν να παροπλιστούν αυτοί που αλλιεύουν παράκτια. Θεωρώ λοιπόν ότι αν γίνει αφο, παροπλισμό, συγγνώμη, θα πρέπει να μας αφορά όλους, όλους τους τόλους και θα πρέπει να έχουμε διακρίσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι ότι οι παραχωρήσει των ποσοστώσεων, το να λέμε ότι οι παραχωρήσει των ποσοστώσεων θα είναι καλό για τη βιωσιμότητα κτλ. αυτό ω επιχείρημα δεν στέκει. Δεν στέκει. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε συζήτηση, είναι καλό να συζητάμε για τις απορρίψει κλπ. Αλλά κανείς νομίζω δεν μπορεί να πει ειλικρινά ότι εγώ είμαι κατά του περιορισμού των απορρίψεων. Όλοι είμαστε υπέρ του περιορισμού των απορρίψεων και χάρηκα που η Κομισιόν το είπε σήμερα το πρωί. Είπε ότι θα πρέπει να γίνονται τεχνικέ και οικονομικέ αξιολογήσει, το οποίο σημαίνει ότι τα, πλέα ότι τα, συγγνώμη, λιώματα θα πρέπει να ρίχνονται στη θάλασσα με το σωστό τρόπο και θα πρέπει να δούμε τι οικονομικές επιπτώσεις έχουν όλα αυτά. Εντάξει, για τι απορρίψει λοιπόν ξαναλέω συμφωνούμε όλοι, όμω θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλο τρόπο, η κατάλληλη συντογή με την οποία θα πρέπει να, γίνονται, να γίνει ο περιορισμό των απορρίψεων και να έχουμε και τι κατάλληλε τεχνικέ προδιαγραφέ και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τα δίχτυα και άλλα τεχνικά ζητήματα που θα μα επιτρέψουν να το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν γίνεται να στείλουμε ας πούμε ένα SMS ή ένα email στα σκάφη και να λέμε κοιτάξτε να δείτε αυτό το αλίευμα ξέρω το τάδε ψάρι έξω το θάλασσα. Αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχουμε ας πούμε μεγαλύτερα δίχτυα για συγκεκριμένα είδη ψαριών. Και σε σχέση τώρα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ως σύσταση νομίζω ότι δεν γίνεται να το βελτιώσουμε και τόσο πολύ αυτό και ο κύριος ε, Στίβενς νομίζω είχε πει κάποια πράγματα για την κοινή οργάνωση αγοράς. Αν γίνεται να φτάσουμε μέχρι το 2012 δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό το πράγμα αν αυτό είναι εφικτό, αλλιώς θα πρέπει να πάμε αργότερα, πούμε, το 2013-2014 και μετά. Ευχαριστώ κύριο Σφάκτο. Um, uh, Ενδιαφέρουσα υπόψη των Ιρλανδών και εγώ άκουσα τις απόψεις διαφορών μελών εδώ της Επιτροπής. Βεβαίω, εμείς είμαστε νομικοί όλοι. Είμαστε όμως ε, νομοθέτες μέσω της απόφασης. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο ισχύων νόμος απέτυχε όσον αφορά τους στόχους του. Το είπε και η Κομισιόν εξάλλου. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Και όπως είπε και ο κύριος από την Κομισιόν, εμείς έχουμε ευκαιρία ως νομοθέτες να κάνουμε κάτι σωστό εδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά να κάνουμε κάτι το σωστό όπως έλεγα προηγουμένως. Ξεκίνησαν συζητήσεις για αυτά τα θέματα σε κάποια φόρουμ πριν από κάποιο καιρό. Μιλήσαμε για την περιφερειοποίηση, για την χάραξη αλληλευτικής πολιτικής που θα είναι αποτελεσματική, αποκέντρωση σε μέγιστο επίπεδο. Αλλά είχαμε τόσες πολλές προτάσεις σε κεντρικό επίπεδο που δεν είχε μείνει και τίποτα να αποκεντροποιήσουμε εκτός από αυτές τις ε, υποχρεωτικές τέλο πάντων ε, ε, παραχωρήσεις και τις ποσοστώσεις. Τώρα για τις απορρίψεις. Νομίζω ότι η Κομισιόν είναι κατά των απορρίψεων σαφώς αλλά πριν από δύο εβδομάδες είδαμε προτάσεις της Κομισιόν για ποσοστός οι οποίες θα αυξήσουν τις απορρίψεις. Πρέπει λοιπόν τώρα η Κομισιόν να μας αποδείξει με τις επερχόμενες προτάσεις της ότι πράγματι θέλει να κάνει κάτι εδώ σε αυτόν τον τομέα και ότι έχει την βούληση να το κάνει Και να πούμε ότι εντάξει έχουμε από αποκέντρωση τα θέματα νομικά, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν με πείθηκε τόσο αυτό το επιχείρημα. Και δεν πιστεύω και τόσο σε αυτό που λέει η Κομισιόν ότι οι νομικοί σύμβουλοι τέλο πάντων τις δένουν τα χέρια κατά κάποιο τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φαρέρα και με τα σχόλιά του για τα όρια Και η Κομισιόν νομίζω έχει παραδεχτεί ότι το όριο των 12 μιλίων δεν είχε την κατάλληλη διαχείριση και ότι αυτός ο λόγος ο αυτός θα ήταν ο λόγος για να εξετάσουμε προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν εδώ τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν. Τι είπε και ο κύριος Φαρά, νομίζω 200 μίλια, εντάξει. Αυτό θα ήταν πολύ καλό, αλλά βεβαίως θα πρέπει να αυξήσουμε τα όρια. Και τελευταία φορά που το είχαμε συζητήσει εδώ, είχα εκφράσει την ίδια άποψη. Τώρα νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να έχουμε και αυτό που μας λείπει υπό την τωρινή ελευθερική πολιτική είναι το να πάμε σε μια κατάσταση όπου αυτοί που έχουν να κερδίσουν περισσότερο από τη διατήρηση, δηλαδή αλληλεί, έχουν ένα κίνητρο, δηλαδή ότι οι ίδιοι θα επωφεληθούν μακροπρόθεσμα από τα δικά τους μέτρα διατήρησης και τις βασικές προδιαγραφές και απαιτήσει. Όμω αυτό δεν βλέπω πώ θα το πετύχουμε αν πούμε ότι έχουμε τέλο πάντων μια κοινή θάλασσα η οποία είναι προσβάσιμη σε όλου, σε ίση βάση δηλαδή, και ότι η αποκέντρωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα. Νομίζω ότι στο μέγιστο θα πρέπει να εφαρμόζεται η αποκέντρωση. Εμείς θα το επιθυμούσαμε αυτό οπωσδήποτε, και θα θέλαμε ομάδες αλευτικών χωρών να διαχειρίζονται τις δικές τους θάλασσες για δικό τους μακροπρόθεσμο όφελος. Ευχαριστώ. Ε, τέλος κυρία Τράουτμαν και κλείνουμε τη λίστα των ομιλητών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να έρθω σε κάποιες πτυχές οικονομικές ε, για να μην ξαναπώ αυτά που είπαν πολύ καλά συνάδελφοι. Όπως είπε η κυρία Λέβιν και, και ο προηγούμενος, ο προναλήσα συνάδελφος, επίσης, εμείς θα πρέπει να προσέξουμε ότι τα... αυτό που είναι σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τους πόρους αυτό, η αλληλευτικοί πόροι και η προστασία τους είναι το α και το μέα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να προστατεύσουμε τον τομέα λοιπόν, αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι και ακριβείς όσον αφορά τις οικονομικές πτυχές. Στη χώρα μου για παράδειγμα σήμερα είναι δύσκολο να διατηρηθούν, ε, να λειτουργήσουν ορισμένες ε, εταιρείε, να κρατήσουν τους ε, εργαζόμενούς τους υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Απ' τη μια μιλάει κανείς για διατήρηση των πόρων, ε, διαλέει τις ε, ποσοστώσεις όσον αφορά την αλληλεία, ατομικές άδειες κτλ. και μεταφέρσιμες, αλλά δεν προχωράει όσο πρέπει στην ανάλυση για τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Ε, για την κερδοσκοπία φέρει πίν, που μπορεί να γίνει γύρω από τον αλληλευτικό τομέα. Επίσης, οι επιβαρύνσεις στις εταιρείες μπορεί να υπάρξουν και κυρίω όταν μιλάμε το θέμα των απορρίψεων των αλλιευμάτων. Εδώ βλέπω πολλά ερωτηματικά να τίθενται. Έχουν να κάνουμε με τα λέματα τα οποία είναι πολύ μικρά, που χρησιμοποιούνται για να γίνονται ε, άλευρα για ζώα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, Γίνεται, είναι, έχουμε εδώ μια επιλογή οικονομική, πρέπει κανείς να αποφασίσει πώς ακριβώς θα γίνει η χρήση και με ποιο τρόπο. Τι γίνεται επίση με το θέμα όταν έχουμε να κάνουμε με ε, αλλιέματα τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα. Μήπως θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τα διάφορα συστήματα επιλογών, επιλογών αυτό που εφαρμόζεται στις αλευτικές εταιρείες. Να δει κανείς το θέμα που των επιπτώσεων των συνθηκών εργασίας και γενικότερα τις οικονομικές συνθήκες για τις εταιρείε. Όλα αυτά σας ανέφερα έτσι γρήγορα είναι στοιχεία πάνω στα οποία θα πρέπει να προβληματιστούμε να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να κάνουμε τον τομέα αυτό πολύ πιο υπεύθυνο. Τώρα, αν κανείς παρατηρήσει στον συνδυασμό σε σχέση με τους προσανατολισμούς που έχουμε μπροστά μας για τις ποσοστώσεις που μπορούν να μεταφερθούν κτλ. Τι διαπιστώνει κανείς. Έχουμε ένα θέμα το οποίο ανέφεραν συνάδελφοι που αναφέρθηκαν στο θέμα της περιφερειοποίησης αλλά έχουμε όπως ελέγχθη τον κίνδυνο να υπάρχει συγκεντρωτισμός Έχουμε από τη μια στόλους που είναι δραστηριοποιημένοι σε ένα ε, χώρο, αλλά έχουμε και αυτό που θέλουμε να υποστηρίξουμε, δηλαδή την παράκτη αλία. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τη διάσταση αυτή που έχει να κάνει με τις παράκτιες ζώνες. Έχουμε μετά και την ε, ε που γίνεται, αεραστεχνική θα λέγαμε αλληλεία, όπου δεν υπάρχουν οι ίδιοι έλεγχοι, δεν υπάρχουν οι ίδιες υποχρεώσεις που εφαρμόζει κανείς ε, στην επαγγελματική αλληλεία. Αυτά σαν προβληματισμό ήθελα να θέσω στο διάλογο που έχουμε κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια σύντομα λέει Πρόεδρος. Προσωπικά με απογοήτευσε πολύ μεταρρύθμιση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι, όπως είπε και κάποιος, την παρουσίασε σε σχέση με κάποιες μικροπροσαρμογές ή επαναχωρήσεις σε σχέση με παλαιότερες θέσεις τους. Νομίζω ότι οι συζητήσεις που είχαν με χώρες μέλη και επαγγελματικού φορείς σε σχέση με τα διάφορα στοιχεία της μεταρρύθμισης Αυτά δεν έγιναν δεκτά και αποσύρθηκαν πριν μπουν σε μια ουσιώδη συζήτηση. Ελευθερή πρόσβαση και άλλα στοιχεία, γιατί εδώ έγιναν δεκτά τα status quo διαφόρων θεμάτων χωρίς να τα έχει συζητήσει κανείς, να τα έχει υποστηρίξει. Παραχώρησαν λοιπόν σε σχέση με πολλά θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν συζητήσει και να επαναπροσδιορίσει Παίρνω προηγούμενο σε αυτό το οποίο η Επιτροπή ό,τι θεωρεί ότι είναι τα καινούργια στοιχεία τη ε, μεγάλη μεταρρύθμιση, δηλαδή είναι αυτή η περιφερειοποίηση όπω ορίζεται στο άρθρο 4, εκεί που λέει ότι θα οριστούν οι αρμοδιότητε σε κάθε επίπεδο, όμω τώρα μα φαίνεται ότι είναι κενό περιεχομένο. Οπότε ε, έχουμε αυτό το στοιχείο της ε, νομική βάση όπου δεν μα πείθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μα εξηγήσει πώ προβλέπει ότι στο μέλλον θα λάβει κάποιο είδου ε, σάρκα και οστά αυτή η περιφερειοποίηση για να μην είναι κάτι κενό περιεχομένο οπότε παρακαλώ τι είπε ο κ. Στίβενσον να το λάβουμε υπόψη μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα το, το τι γίνεται με την συνθήκη, τι γίνεται με διαχείριση και λέει λέει για τη διαχείριση, λέει για την ε, διατήρηση των ε, πόρων. Θα πρέπει να δούμε όλα αυτά, από τι, τι, τι, μορφή έχουν λάβει, για να δούμε τι θα γίνει με την περιφερειοποίηση. Οπότε όλα αυτά έχουν σχέση και με αυτό το οποίο εσείς μας είπατε, κάτι το οποίο αφορά ε, τα πολιετή προγράμματα. Τι γίνεται. Ε, τι σχέση έχει αυτό με την περιφερειοποίηση όταν τα περισσότερα βασικά στοιχεία του πολιετούς προγράμματος είναι προκαθορισμένα. Οι απορρίψεις ε, <clears throat> τα των ελληνικών πόρων. Οπότε, εάν το έχει προκαθορίσει η Επιτροπή, τι γίνεται με τους πόρους και την ε, απόδοση, τι γίνεται με τις απορρίψεις, τότε τι θα τα κάνουμε τα πολιετή προγράμματα επίσης. είναι για την αλία αυτά τα προγράμματα γιατί ο ορισμός των πολιτών προγραμμάτων δεν λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της ιδιομορφίας της αλίας. Λάβετε επίσης υπόψη τι γίνεται όσον αφορά τη μεγίστη βιώσιμη απόδειξη. Απο, α, απόρριψη. Σήμερα αυτό το οποίο έχουμε ως βιώσιμη απόδοση πρόκειται να είναι εφικτό το 2015. Βρείτε έναν ορισμό, περιχαρακώστε κάπου την έννοια αυτή, ούτως ώστε αυτό να στέκει. Επίσης, νομίζω ότι σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις υπολείπεται η τωρινή. Για τις ποσοστώσεις επίσης. Έχουμε εδώ αυτό το οποίο θέλουμε, μείωση δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος το να υπάρχει σύστημα εκούσιο. Τι να κάνουμε, να μην αυτό το σύστημα όπως είναι. Τότε δεν κάνουμε τίποτα. Και πάμε για συρρήκνωση του στόλου επομένω. Όμως δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τις ποσοστώσεις. Και από την άλλη μεριά σας ρωτώ, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται στη χώρα σας. Αμφιβάλλω ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη χώρα. Κανένας ψαράς πουθενά δεν έχει ελεύθερη πρόσβαση. Πού τα βρήκατε αυτά. Μόνο όσοι έχουν την άδεια. Οι άλλοι δεν επιτρέπεται να ψαρέψουν. Να μην λέμε λοιπόν ότι, ότι τώρα βρήκαμε το αυγό του Κολόμβου και βρήκαμε τη λύση. Όχι. Όμως έτσι δεν αλλάζει το σύστημα. Για να αλλάζει το σύστημα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως ότι έχει αποδώσει το σύστημα, έχει οικονομικό ενδιαφέρον. Έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο. Αν δεν έχετε να προτείνετε κάτι, νομίζω ότι όπως έχει σήμερα το σύστημα είναι το καλύτερο για να πετύχουμε του στόχους που όλοι θέλουμε. Κύριε Πένια, θέλετε το λόγο, δεν ξέρω. Παρακαλώ, παρακαλώ να είσαστε σύντομος. Άλλωστε, όλα αυτά τα θέματα θα ξαναζητηθούν και αναλυτικά ένα προς ένα. Όμως, ας αφήσουμε μισή ώρα ούτως ώστε οι άλλοι δύο συνάδελφοι να μιλήσουν για τα θέματά τους. Έχουμε τις ανακοινώσεις των συναδέλφων. Το θέμα θα ξαναζητηθεί σε όλες μας τις συναντήσεις. Ας δούμε επομένως τα θέματα όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα από είπε κύριε Ρόντος. Παρακαλώ πέντε λεπτά μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά για, μέσα σε πέντε λεπτά και. Το θέμα του κυρίου Ντέβις ε, είναι κάτι που θα με απασχολήσει. Τέλος πάντων ε, δεν θα απαντήσω. Θα απαντήσω για να καλύψω ελπίζω όλου και όχι εσένα ένα από του ε, ε, ερωτήσαντε. Όσον αφορά τι εξωτερικέ εκθέσει σα, διαβεβαιώ ότι με το καινούριο πρόγραμμα θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα, ούτω ώστε να μην έχουμε επικαλύψει όσον αφορά τι επιστημονικέ εκθέσει. Και επίση έχουμε την πρόταση του Νοεμβρίου, ούτω ώστε εκεί που θέλουμε να έχουμε χρηματοδότηση θα πρέπει να δούμε ότι ένας από τους τομείς που θέλουμε να βοηθήσουμε είναι η προετοιμασία των επιστημονικών εκθέσεων. Δεν έχουμε το χρόνο. Όμως, να τα ξαναπούμε όταν θέλετε. Ευχαρίστω να έρθω να σας τα εξηγήσω, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε οπωσδήποτε είναι να αυξηθεί η πρικοδότηση παρά το ότι δεν είναι το μόνο μας πρόβλημα αυτό. Τώρα, κάποιοι που έλαβαν το λόγο είπαν ότι δεν κάνουμε τίποτα για την ε, αλία μικρής κλίμακας. Υπάρχουν εδώ δύο σημαντικά στοιχεία. Γιατί έχουμε τη διαδικασία της διαβούλευσης. Πολλά είπαμε στην, ε, στην πράσινη βίβλο. Αυτά όλα ήταν αποτέλεσμα, όπως είναι λογικό, αποτέλεσμα της διαβούλευσης. και να λάβουμε υπόψη τι έχει γίνει όσον αφορά την αλία μικρής κλίμακας. Δεν υπήρξε ομοφωνία γύρω από την πρόταση της Κομισιόν για ε, καινούριο καθεστώς διαχείρισης χωριστό. Το είπαμε, στην Πράσινη Βίβλο δεν υπήρξε όμως συμφωνία. Τα 12 μίλια ε, ό,τι είχαμε προτείνει γενικά δεν έτυχε ομοφωνίας. Ούτε σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης. Οπότε, παρακαλώ, αναμείνετε στο ακουστικό σας για να δείτε την πρότασή μας για την χρηματοδότηση. Γιατί εκεί θα προκύψει πολύ πιο ξεκάθαρα το τι σας προτείνουμε για την αλληλεία μικρής κλίμακας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο όσον αφορά ε, αυτό που ρωτά το Κοινοβούλιο, όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση και θα πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί κάτι σαφώς όταν μιλούμε για αυτού του είδους της μεταβιβάσιμης άδειας αλίας. Μα το έχουμε πει. δεν πρόκειται για τίτλους κυριότητος. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο είδους δικαιώματα, δικαιωμάτων. Είναι... Δεν είναι με τίποτα ιδιωτικοποίηση. Τα κράτη-μέλη θα χορηγήσουν τις άδειε όπου κρίνουν. Τα δε 12 μίλια. Δεν είναι παρέκκληση ή κανόνας. Δεν είμαι νομικός. Αλλά οι νομικοί μας έχουν αναφέρει ότι καταρχήν η αρχή της ελεύθερης πρόσβασης θα πρέπει να τηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και η αρχή αυτή είναι η βάση μας. Όμως έχουμε τις δύο παρεκκλήσεις. Πρώτον, τα 12 μίλια είναι μια παρέκκληση περιορισμένη. Παρέκκληση της ελεύθερης πρόσβασης. Άλλη παρέκκληση αυτές οι υπεράκτιες περιοχές. Εκεί έχουμε ε, άρθρο στη συνθήκη, συμπάθητα δεν θυμάμαι ποιο είναι, και εκεί επιτρέπεται η θετική διάκριση λόγω των ειδικών συνθήκων αυτών των περιοχών, των υπερακτίων περιοχών. Αζόρες, Κανάρια, Μαδέρα το άρθρο αυτό της συνθήκης ορίζει ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια μεταχείριση. Τώρα, γιατί με αυτές οι μεταφορές είναι υποχρεωτικές, το είπα και το παραλαμβάνω. Αν δεν ήταν υποχρεωτικές, δεν θα άλλαζε τίποτα. Θα μέναμε στα σημερινά. Δηλαδή, θα είχαμε συνέχεια υπεραλίευση. Αυτά όλα το δοκιμάσαμε. Αυτά και άλλα πολλά, πολλά ε, χρήματα από το Δημόσιο Κορβανά για, την, για τον παροπλισμό. Δεν κάνουμε τίποτα σήμερα όσον αφορά την υπεραλήψη. Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και τώρα, σε σχέση με τις ρήτρε διαφύλαξης, με το θα, ότι θα πρέπει ό,τι σύστημα κάνουμε να είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο σχέση με αυτά που θέλει να κάνει η Επίτροπος, γιατί υπάρχουν οι νομικές γνωμοδοτήσεις. Έχω να σας πω το ίδιο επιχείρημα που είπαμε και προηγουμένως, αλλά με θετική διατύπωση. Δικαιώματα μεταβιβάσιμα, με κάποιες ρήτρε διαφύλαξης. Οι νομικοί θεωρούν ότι αυτό είναι συμβατό με την συνθήκη. Είδατε δεν είναι μόνο καλά, κακά μαντάτα αυτά που μας φέρουν οι νομικοί, μα δεν είναι και τίποτα καλό. Όσον αφορά τώρα τις απορρίψεις, γιατί περιοριζόμαστε μόνο σε μερικά λίγα εμπορικά είδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να απορρίψει μέσα σε μια μέρα όλες τις απορρίψεις. Το έχουν κάνει αυτό κάποιες χώρες. Είναι γνωστό ότι έχουν πετύχει. Το πώς το κάνουν τώρα. Λίγο-λίγο προσέθεταν στον κατάλογο ήδη ψαριών. Εμείς εδώ θα μπορούσαμε ναι, να πατήσουμε γκάζι και να τα κάνουμε όλα γρήγορα. Θέλουμε όμως παρόλα αυτά να είναι βαθμιαία η ρύθμιση. ξεκινούμε με τα πιο εύκολα. Όπου είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το νέο καθεστώ για τι απορρίψει. Για τα βασικά είδη, βασικά ψάρια. Βαθμία και στην πρόταση υπάρχει επίσης ένα άρθρο που προβλέπει το ότι μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα είδη σε αυτή την λίστα της αγόρευσης. Ευελιξία βαθμία ρύθμιση και μπορούμε, λέει ξανά ο μιλητή, να προσθέσουμε και άλλα είδη. Και είναι δύσκολο να προδικάσουμε το πού θα καταλήξει αυτό το καθεστώ. Όμω εμεί θα συγκροτήσουμε το μηχανισμό ούτω ώστε να υπάρχουν δυνατότητε ε, κάποια στιγμή κάπου να καταλήξουμε τώρα. Γιατί δεν ακολουθούμε το νορβηγικό μοντέλο. Ότι δηλαδή το σύστημα ελέγχου θα χρηματοδοτείται από τα είδη τα οποία δεν απορρίπτονται. Το μελετήσαμε βεβαίω το νορβηγικό μοντέλο. Όμω δεν το αγκαλιάσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι πρόκειται για μια μικρή χώρα με λίγο κόσμο. Εύκολα έχει κάνει τη διαχείριση. Όμως, αν εμείς προσπαθήσουμε αυτά να τα εφαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι πάρα πολύ περιπλοκό και δεν νομίζω ότι αυτό για πρακτικούς λόγους τώρα είναι εφικτό. Έχουμε πάρα πολλούς λιμένες εκφόρτωσης στην Ευρώπη. Επομένως δεν είναι το θέμα φιλοσοφικό. Ε, λέει ο μιλητής η Νορβηγία είναι μικρή χώρα με λίγο κόσμο και εδώ θα ήταν πιο πολύπλοκο. Οπότε, αν γινόταν θα το κάναμε γιατί δεν θεσπίζουμε κανόνες ούτως ώστε τα κρατημέλη να μπορούν αυτά τα ε, με τα βιβάσιμα δικαιώματα να τα χορηγούν, να τα εκχωρούν σε αυτούς που συμπεριφέρονται σωστά. Μα υπάρχει κάποια παράδοση. Τα κράτη-μέλη ε, καθορίζουν και διανέμουν τις ποσοστώσεις. Εμείς το σεβόμαστε. Και είπαμε ότι στην πρότασή μας δεν υποχρεώνουμε, δεν περιορίζουμε κανένα. Τα κράτη-μέλη να κάνουν επομένως αυτήν την διανομή. Και με κάποια ενεργή πολιτική να αμείβουν το ΣΥΠΗΝ αυτούς που έχουν σωστή συμπεριφορά. Hemos que hay que preservar de dejar esto al Estado miembro, como ha sido hasta ahora. Eh, vamos a ver, la, la cuestión de la... Παρακάτω η κοινωνική πτυχή που είπατε ότι δεν προβάλλεται και πάρα πολύ να κάνουμε εδώ πέρα κάποια διάκριση. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Επί τη βάση της κοινή πολιτικής δεν μπορούμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Άλλη νομική βάση, άλλη αρμοδιότητα, όλος διαφορετική. Άρα δεν μπορούμε άμεσα να νομοθετήσουμε. Αυτό σημαίνει βέβαια δεν μας απασχολεί το κοινωνικό θέμα, φυσικά και μας ε, απασχολεί. Και έχουμε εδώ τώρα δύο ή τρία βασικά στοιχεία. Το ότι μας απασχολεί σαφώς η αλληλεία μικρής κλίμακας, γιατί έχει κοινωνική διάσταση, σύμφωνη. Αλλά αυτό το θέμα με το ε, μεταβιβάσιμων αδειών έχουν, έχει κάποια θετικά. Όπου εφαρμόστηκε, απέδωσε. Και έτσι είχαμε καλύτερη μισθολογική πολιτική. Ο κλάδος. Δυστυχώς δεν προσφέρει δουλειά ελκυστική για τους νέους. Δηλαδή το να μπαρκάρουν και να δουλέψουν πάνω στα ελευτικά. Όμως, όπου εφαρμόστηκε η εν λόγω πολιτική, οδήγησε σε καλύτερα μεροκάματα και άρα έκανε πιο ελκυστικά τα ελευτικά σκάφη. Τη δουλειά πως τα ελκυστικά σκάφη για τους νέους. Άρα, να, γεωνική επιτυχία. Και θα τα δείτε όταν έρθει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Δεν υπάρχει τώρα χρόνος να σας τα πω. Εάν μου επιτρέπετε όμως κυρία Πρόεδρε, να αναβληθεί η σχετική συζήτηση όποτε μπορέσουμε. Το Δεκέμβριο, όταν έρθει η ώρα. Άλλο. Γιατί δεν νομοθετούμε όσον αφορά την αηλία ως σπορ. Ήδη αυτά τα συζητήσαμε. Ήδη τα συζητήσαμε σε σχέση με τον ελεγκτικό κανονισμό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αμφιλεγόμενος και είπαμε ότι σε περίπτωση που η Ελία e ως πορ αναβαθμιστεί ή όσον αφορά τους πόρους έχει επιπτώσεις, τότε θα ληφθούν μέτρα σε κοινωνικό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε με τίποτε να ρυθμίσουμε εδώ από τις Βρυξέλλες την αλία ως σπορ. Είναι θέμα κρατών μελών. Εκεί που έπρεπε νομοθετήσαμε. Να, και ο κανονισμός για τη Μεσόγειο. Τα ξέρετε. Εκεί, για κάποιους τρόπους αλίας παρα, ε, ε, ε, επαγγελματικούς υπάρχει απαγόρευση στη χρήση τους από τους ε, αλληλείς σπόρτσμεν, ας πούμε. Ή είπαμε τώρα ότι θα πρέπει να... Παρακαλώ ολοκληρώστε, λέει Πρόεδρος. Το τελευταίο, τελευταίο, τελευταίο. Κύριε Πρόεδρε, σας απαντώ με ερώτηση. Εάν θέλετε να προχωρήσουμε περισσότερο για την περιφερειοποίηση, για πέστε μας, θέλετε η μεγίστη απόδοση να κανονιστεί σε επίπεδο περιφερειακό. Είσαστε εσείς οι συνομοθέτες με το Συμβούλιο. Εσείς τα βασικότερα μέτρα θα τα υιοθετήσετε. Αποφασίστε ό,τι θέλετε. Εσείς άρα θεωρείτε η μεγίστη βιώσιμη απόδοση θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νομοθεσία. Όχι, λοιπόν, δεν θεωρούμε νέο, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και θεωρούμε ότι αυτό δεν αντιβαίνει στην περιφερειοποίηση. Ακριβώ όπω τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι όπω τα λέτε εσεί, τα γυρίζετε και το κάνετε να αντιβαίνει. Αλλά δεν είναι έτσι, λέμε εμεί, λέει η Πρόεδρο. Τώρα στη συνέχεια, εάν συμφωνείτε, να δώσουμε για 15 λεπτά στον καθένα από τους ε, αγορητές και μετά στην Κομισιόν χωρίς ε, παρεμβάσεις για τις αγορές εξωτερική πολιτική. Εάν λάβετε το λόγο δεν μπορούμε. Θα πρέπει το θέμα να το αναβάλουμε. Pero les propongo que como primera medida, dado que están aquí, está aquí la comisión, hoy actuemos así y en el futuro tendremos más tiempo para los demás de... Άρα θα πούμε αυτά και στο μέλλον να δώσουμε περισσότερο χρόνο για την ίδια ζήτηση. Κύριε Στίβενς, έχετε το λόγο. Very much, Chairman. On the timetable for the... Για το χροδιάγραμμα. Εγώ σας προτείνω το ίδιο για την κοινή οργάνωση αγορών. Να δούμε τι θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου. Τότε να τα πούμε περισσότερο όσον αφορά. Και έχουμε 25 και 24 και 25 τον Ιανουάριο έχουμε μια ακρόαση, συνακρόαση. Επίσης έχουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια στις 29 Φρουαρίου. Τότε θα σας πω Μάλλον όχι, θα μπορέσω αφού τα συζητήσουμε τέλο Μαρτίου να σα παραλυθεί το τελικό μου κείμενο και να έχουμε και, την προθεσμία για τι τροπολογίε 24 και 25 Απριλίου. Και ψήφιση 30 Μαΐου. Οπότε θα κατέβει το θέμα στην Ολομέλεια, όπως και ο Γερόντος, στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Τα βασικότερα σημεία τρόπου που θα να συζητήσουμε είναι πώς η κοινή οργάνωση αγοράς θα βοηθήσει στη βιώσιμη ε, αλία. Να μήψουμε τους καλούς μαθητές, να τιμωρήσουμε τους κακούς, να έχει περισσότερη συνοχή η αγορά, να έχουμε ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, να αντιμετωπίσουμε την προβλεψιμότητα της αγοράς, Βεβαίως όλα αυτά με δεδομένο το ότι αυξάνεται η ζήτηση για ψάρια στην Ευρώπη. Αλλά να δούμε, να εξετάσουμε τι ζητούν οι καταναλωτές. Από την άλλη μεριά να αποφύγουμε την πολυνομία και την γραφειοκρατία. Να κάνουμε απλούστευση. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Τα βασικά σημεία που θέλουμε να εντοπίσουμε, ελπίζω, με τη βοήθεια ειδικών ή με τη βοήθεια της διαβούλευσης. Ο επόμενος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κομισιόν. Ακριβώς όπως είπατε, αυτό είναι το μήμα της γενικότερης μεταρρύθμισης. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πώς γίνεται η παραγωγή. Οπότε να δούμε πώς είναι οργανωμένη η αγορά και να δούμε τη διεθνή διάσταση. Όπως είπε ο κ. Στίβενσον, ένα από τα βασικά σημεία στην οργάνωση της αγοράς είναι ότι πάσχει από γραφειοκρατία. Να γίνει απλούστευση, να αντιμετωπίσουμε την περιπλοκότητα, να δούμε εκεί οι οικονομικοί παράγοντες και η παρέμβαση πώς θα λειτουργήσουν και τι θα γίνει με την ενδικατοθεσία. Απλούστευση πρώτον. Μείωση νομοθετημάτων. Τέσσερις κανονισμοί, τρεις εφαρμοστικοί, να έχουμε έναν με συναπόφαση και τέσσερις ε, εφαρμοστικέ πράξεις και κατανάθεση πράξη. Απλούστευση θα είναι ευξημένες ευθύνες των ε, εμπλεκομένων να μειωθούν, να μειωθούν οι, υποχρεώ, οι περιπτώσεις υποχρέωσης ε, κοινοποίησης, και γενικότερα και στο χρηματοδοτικό μέσο απλούστευση να έχουμε ένα και μόνο μέσο χρηματοδότησης. Άλλο. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των εμπλεκομένων. Ισχυρότερες οργανώσεις παραγωγών με περισσότερες ευθύνες. Ενίσχυση των οργανώσεων όλων των εμπλεκομένων μέσω συνεργασίας με αυτές αναγνώριση, υποστήριξη διεθνών πρωτοβουλειών. και να δράσουμε με οικονομική ευφυΐα ούτως ώστε να ξέρουμε καλύτερα, να έχουμε περισσότερες απόψεις για το τι γίνεται στην αγορά και όσον αφορά την οικονομική λειτουργία της αγοράς. Και έτσι να είναι πιο σωστή η αντίδραση και η παρέμβαση στις αγορές. Τρίτο στοιχείο, η θέσπιση, τέλο πάντων η επινόηση νέας λογικής παρέμβαση στην αγορά. Λοιπόν, να γίνει μια πρώτη αναθεώρηση των προτύπων των προϊόντων. Και άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο προγραμματισμός και το marketing για τις παραγωγές. Για την παραγωγή μάλλον, τόσο ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την παραγωγή. Να δούμε τι πραγματικά γίνεται. περιορίζεται κανεί να ασχοληθεί με, το, με τον πρώτο κρίκο τη παραγωγή ή όχι. Να α πούμε, οι να ασχολούνται μόνο με το να πιάνουν τα ψάρια ή να φτάνει η ασχολία του, η ευθύνη του μέχρι να φτάσει στο πιάτο του καταναλωτή, ούτω ώστε και έτσι να ωφελείται περισσότερο παραγωγό, να υπάρχει δηλαδή περισσότερη σύνδεση παραγωγή με κατανάλωση. Τώρα. Ε, ο μηχανισμό παρέμβαση. Και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε αλλαγή, αναστολή υποστήριξης, βάσει της λογικής του να περιορίσουμε τη διασπάθηση των τροφίμων. Ενιαίο μηχανισμό αποθήκευσης και αποθεματοποίησης. Και έτσι να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την παραγωγή και το μάρκετινγκ, τη θέση σε εμπορία. Όταν δεν προσφέρεται η χρονική στιγμή για θέση εμπορία, τότε να πηγαίνουμε σε αυτήν την αποθήκευση, αποθεματοποίηση. Και να δούμε όμως και αυτό από εδώ, αυτό τι, τι μπορεί να βγει. Αναβάθμιση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών και τέλος η δικαιοτόθεση για την υπεύθυνη κατανάλωση. Υποχρεωτικά να παρέχονται πληροφορίε επί του προϊόντος. Και με τα μεταποιημένα και στην κονσέρβα. Να υπάρχει ακρίβεια, ξεκάθαρη πληροφορία, προέλευση των προϊόντων ανιχνευσιμότητα, δείχνει λασιμότητα. Να ξέρει ο καταναλωτής από πού προέρχεται το προϊόν. Από το δίχτυ μέχρι το πιάτο. Πληροφορία επίση για την ελίευση, ημερομηνία, ε, απόψυξη, ε, πότε αν έχει γίνει και επίσης ε, ένα πλαίσιο για θελούσια υπαρχή πληροφοριών με κάθε επιφύλαξη των όσων ορίζει ο νόμος. Και έτσι να είναι δυνατή η διατύπωση θεμητών αξιώσεων για το προϊόν. Και ο καταναλωτής να ξέρει καλύτερα τι παρήχθη, τι καταναλώνει και όπου αξίζει ένα προϊόν να πληρώνει και κάτι παραπάνω καταναλωτής. Ε, Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο σημείο. Ανακοίνωση εξωτερικής πολιτικής. κυρία Λεβίν. Το σημείο 16, εξωτερική διάσταση κίνηση ανοιχτή πολιτικής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε οριστικό χρονοδιάγραμμα. Αλλά θα έχουμε έγγραφο εργασία. Δύο. Και αυτό που εξετάζουμε εδώ είναι οι συμφωνίες αλληλείας εταιρικής σχέσης που θα είναι βιώσιμες, για βιώσιμη αλληλεία δηλαδή, και οι προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της απόδοσης. Να υπογραμμίσουμε επίση και τις ρυθμίσεις με τρίτες χώρες και συμφωνίες κοινωνικού πλαισίου όπως επίσης η διαφάνεια σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Αυτά θα συζητηθούν στους επόμενους μήνες. Να μου πει τώρα η Κομισιόν την πρότασή της. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Τρίτο σημείο που έχει να κάνει περισσότερο με προθέσεις πολιτικής και δηλώσεις και όχι με νομικά στοιχεία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Πρώτο στοιχείο με την παρουσία των στόλων μας στους ωκεανούς. 24% προέρχονται από τα λιεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλες θάλασσες. Πρώτο στοιχείο αυτό. Δεύτερο, οργάνωση αγοράς. Σημαντική επειδή η αγορά μας είναι μεγάλη. Πάνω από τα δύο τρίτα της κατανάλωσης είναι εισαγόμενα. Θεωρούμε λοιπόν να θα πρέπει να δούμε το πώς οι πόροι θα διαχειρίζονται παντού, παγκοσμίω, ώστε να υπάρχει ασφάλεια για όλους τους καταναλωτές. Εξωτερική διάσταση. Καταρχήν έχουμε το Διεθνή Οργανισμό για τη Διαχείριση των αλληλευμάτων. Έχουμε τα όργανα Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών και συμμετείχαμε ως ΕΕ σε όλα τα σώματα. Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος, αλλά είμαστε παρατηρητές σε πολλά από αυτά, ώστε να έχουμε κάποια παρουσία. Είμαστε μεγάλος παίκτης Προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις απόψεις στα RFMOs και να βεβαιωθούμε ότι εισακούονται οι προτάσεις μας και οι απόψεις μας. Το θέμα όμως της βιώσιμης αλληλείας θέλουμε να το αναγάγουμε σε παγκόσμιο. Τα λεπτομέρειες στοιχεία δεν έχουν τόσο σημασία, αλλά 85% των παγκοσμίων αποθεμάτων υπεραλλιεύονται ή αλλιεύονται πλήρω. Οπότε εμείς έχουμε μια διεθνή ευθύνη οι συζητήσεις στα RFMOs να οδηγήσουν σε μια καλύτερη διαχείριση. Οπότε είμαστε πολύ παρόντες στα RFMOs ώστε η βιωσιμότητα και η χρηστή διαχείριση να διασφαλίζονται. Μπορούμε άμεσα να δουλέψουμε στα RFMOs με την παρουσία μας, αλλά και δημερός μιλώντας στους κύριους εταίρους εδώ και συνάπτοντας συμμαχίες, αν θέλετε, και είναι σημαντικό διμερός να έχουμε συμμαχίες με τους μεγάλους παίχτες αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Π.χ. αλία Αγίου. Σημαντικό αυτό, το οποίο συμπιστήσαμε σε ΗΠΑ Πολιτείες και κάναμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας για τα RFMOs. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το εξής. Να βεβαιωθούμε ότι η απόδοση του είναι βέλτιστη, ότι είναι όσο πιο αποδοτικά όσο γίνεται, ότι οι τεχνικές συμβουλές που υπάρχουν βελτιώνονται, να βεβαιωθούμε επίσης ότι τα μέρη τηρούν τις συμφωνίες, ότι υπάρχουν οι τηρούμενες ανθεωρήσεις και ότι για τα RFMOs μελλοντικά θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα της υπερδυνατότητας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα διεθνώς είναι και το FAO των ΗΕ όπου και εκεί είμαστε ενεργώς συμμετέχοντας στις τεχνικές συζητήσεις. Πολύ συχνά είμαστε και πρωταγωνιστές όταν έχουμε να κάνουμε πούμε, συμφωνίες για συγκεκριμένα μέτρα ή θέματα για τα οποία επικυρώσαμε συμφωνίες από τις πρώτους παγκοσμίω. Ένα άλλο στοιχείο είναι η συμφωνία για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοπικιλότητας πέραν εθνικών θέμα αυτό όπου είμαστε μπροστάριδες και να αναφέρω και μια εκδήλωση του χρόνου το Rio Plus 20 20 όπου η Κομισιόν δραματίζει ενεργό ρόλο και προσπαθούμε να προωθήσουμε σημαντικά θέματα. Βλέπω και το ρολόι, ώρα έχει περάσει και όλοι τα έχουν φτύσει. Σε δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι οι διμερείς συμφωνίες όπου θα πρέπει να κοιτάξουμε διάφορα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν με την ιδέα να τα μεταμορφώσουμε σε συμφωνίες βιώσιμης αλληλείας και να περιλάβουμε εδώ διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να αλλάχθουν ώστε να τροποποιήσουμε και, τις, και τα επιστημονικά στοιχεία και να τα προσαρμόσουμε ώστε να μην αντιμετωπίσουμε μόνο το θέμα δηλαδή των αποθεμάτων αλλά και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πρόσβασης από τους εταίρους μας και να πω επί τη ευκαιρία ότι υπάρχει μια επιστημονική βούληση τη μεγιστοποίηση της ε, αλευτικής ε, δυνατότητας μέσω στόλων Και βεβαίως υπάρχει και μία ποσότητα συμπληρωματική η οποία θα μπορούσε να ληφθεί από άλλους. Εμείς το ζητάμε αυτό, αλλά ξέρουμε ότι και άλλα μέρη και αλευτικοί εταίροι το επιζητούν. Δεν βιαζόμαστε όμως. Θέλουμε οι ποσότητες που έχουν ε, συμφωνηθεί να τηρούνται από όλες τις μεριές. Αυτά είναι τα κυρία στοιχεία. Καλύτερη αξιολόγηση της αλληλευτικής ε, δυνατότητας, ενημέρωση σε σχέση με τις ποσότητες οι οποίες παρέχονται σε άλλες χώρες εκτός δηλαδή ΕΕ, αξιολόγηση συνολικής αλληλευτικής δυνατότητας και επίσης βελτίωση της τομεακής συνεργασίας. Ξέρουμε για τα FPS έχουμε δύο στοιχεία σημαντικά. Πρόσβαση και αληφτικά δικαιώματα. Και θέλουμε οι χώρες επίσης να βελτιώσουν τις νομές για τη διαχείριση του τομέα αλίας γενικότερα. Άλλο ένα στοιχείο αυτό δηλαδή. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι τα κονδύλια στοχεύονται σωστά και ότι τα διαθέσιμα χρήματα λαμβάνουν υπόψη τους την αληθική δυνατότητα ή τη δυνατότητα αφομοίωσης των χωρών στις οποίες προορίζονται αυτά τα κονδύλια. Μέχρι τώρα είδαμε ότι αυτό δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικό επειδή υπήρχε η τη δυνατοτητα φωμιεση των χωρων στις οποιες προοριζονται αυτα τα κονδυλια μεχρι τωρα υποχρέωση για εξόφληση έστω και αν τα χρήματα δεν δίδονταν τομεακά. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα πάνε εκεί που θέλουμε να πάνε. Να βεβαιωθούμε δηλαδή ότι θα έχουμε διάκριση μελλοντικά δικαιώματα πρόσβαση αφενός, τεχνική συνεργασία αφετέρου. Άλλα στοιχεία. Στα FPAs η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για πρόσβαση και οι ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες και οι αλληλείς πληρώνουν Θέλουμε όμως να ισορροπήσουμε αυτή την κατάσταση κάπως και να καλέσουμε τους πλειοκτήτες να αναλάβουν μεγαλύτερο τμήμα του κόστους της πρόσβασης. Κάτι το οποίο σε κάποιες θα μας επιτρέψει να κάνουμε καλύτερη χρήση των χρημάτων που δαπανώνται. Τέλος, θα θεσπίσουμε διατάξεις οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την αλία, όμως αφορούν διατάξεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και λένε ότι τέλος πάντων αν κάνουμε αυτή τη συμφωνία την αυτική με την τάδα και την δίνα χώρα θα πρέπει να τηρούνται βεβαίω κάποια βασικά στοιχεία σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όπου θεωρούμε ότι υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων τότε εμεί ε, αναστέλουμε πρωτόκολλα και σταματάμε συμφωνίε. Και βεβαίως προσβλέπουμε και σε συζητήσεις λεπτομερείς μας για, για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τεντιθέρ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι οι εκθέσεις Λοβίν και Στέβενσον παραπροηγούνται επειδή είναι λιγότερο επίμαχα ως θέματα σε σχέση με άλλα θέματα όπως της κυρίας Ρόντος που χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα κάνουμε μια περιτροπή ώστε να μην ε, μένετε εσείς τελευταία και ξεκάρφατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα το απόγευμα σας περιμένω όλους, σχεδόν όλους, σας πάνω στις 3, στην Ακρόαση δηλαδή, για την παράκτη Αλία και την αλία μικρή κλίμακα σήμερα, το απόγευμα στις 3. Σας προσκαλώ να έρθετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.